Possiamo iniziare, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στις συνεδρίες της Επιτροπής μας. Πρώτο σημείο είναι η έγκριση της μερίσιας διάταξης. Αν δεν έχετε σχόλια, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσεις του Προέδρου. Όπως πάντα η συνεδρίασή μας ε, βγαίνει στο διαδίκτυο. Τρίτο σημείο, προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Είναι το τρίτο σημείο, εισηγητής ο Γιάννος Βοητσιετσκόφσκι. Σούλα. Έχουμε λοιπόν ανταλλαγή απόψεων. Η έκθεση παρουσιάστηκε ο κύριος Δεν ακούω τα αγγλικά. Ακούν οι υπόλοιποι. It's okay? Λειτουργεί τώρα. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, όπω έλεγα, περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων, ε, την οποία δεν συζητήσαμε την πρώτη φορά, έκθεση για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Δεύτερη ανταλλαγή απόψεων με στόχο η Επιτροπή μα. να έχει περισσότερα στοιχεία για τη μεταφορά ζώων των ζώων και έτσι θα μπορέσουμε να ενημερωθούμε καλύτερα για το πώς έχει μεταφράσει το ζώνη εντό Ένωσης και να εκπονηθεί καλύτερα η έκθεση πρωτοβουλίας του Αντιπρόεδρου μας κυρίου Βοητσιακόφσκη. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την Κομισιόν, εν συνεχεία τον εισηγητή και μετά θα ακολουθεί η συζήτηση. Επιτροπή. Thank you very much. Good afternoon. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε κάποια γεγονότα και στοιχεία που κατά την άποψή μας είναι πολύ χρήσιμα και θα βοηθήσουν και την δική σας μελλοντική συζήτηση. Έχουμε λοιπόν κάνει ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων, η οποία δείχνει ότι το πραγματικό μέγεθος ε, της μεταφοράς έχει να κάνει με την ε, σφαγή. Θα περάσω κατευθείαν στην παρουσίαση, την οποία φαντάζομαι έχετε λάβει. Αν όχι βέβαια μπορούμε να σας δώσουμε αντίγραφα. Η παρουσίαση αυτή βασίζεται σε δεδομένα από το Traces. Μόνο δηλαδή μεταφορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουμε συμπεριλάβει τα πουλερικά. Βέβαια θα δείτε κάποια για τα πουλερικά σε κάποιες διαφάνειες. Ποια είναι η συνολική εικόνα για όλα τα είδη ζώων. Το 63% όλων των μεταφερόμενων ζώων εντός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφερόμενων ζώων ε, ταξιδεύουν λιγότερο, ε, για διάστημα λιγότερο των 8 ώρων και το 40% όλων των ζώων μεταφέρονται για σφαγή. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι μεταφοράς. Όπως είπα και ευθύς εξ αρχής υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανάλογα με τα είδη. Βλέπετε εδώ στο γράφημα αυτό τη μεταφορά ζών των ζώων, όχι μόνο για σφαγή, το γενικό αριθμό, για οποιοδήποτε λόγο. Βλέπετε λοιπόν σε ποσοστά τα στοιχεία ροζ είναι κάτω από 8 ώρες, ε, πράσινο 8 με 29 ώρες ε, και μπλε πάνω από 29 ώρες διάρκεια της μεταφοράς. Και βλέπετε και τους αριθμούς σε εκατομμύρια, 4,5 εκατομμύρια ε, για τα βοηδή, για, τα, για τους χείρους 29,5, τα πρώτα 4,2, 0,12 τα άλογα και οι μεγαλύτερες ποσότητες 1,216 για τα πουλερικά. προορισμοί. Το μερίδιο των ζώων που μεταφέρονται προς φαγή, το βλέπετε σε αυτό το πίνακα. Από το συνολικό αριθμό, λοιπόν τα 4,5 εκατομμύρια βοηθοί μόνο 500.000, 16% μεταφέρονται για σφαγή. Και εξ αυτών μόνο 0,21 εκατομμύρια μεταφέρονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 8 ωρών. Το ποσοστό του αντίστοιχο είναι 29%. Βλέπω τα περισσότερα ζώα είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια είναι ε, χείρι, 41% για σφαγή και μόνο το 17% ε, εξ αυτών μεταφέρονται για πάνω από 8 ώρες και βλέπετε τα αντίστοιχα νούμερα για πρόβατα, άλογα, για πουλερικά. Δεν έχουμε δεδομένα, μόνο τον συνολικό αριθμό μεταφερόμενων ζώων εντός ένωσης παραλαμβάνω έχουμε. Κάποια πιο αναλυτικά στοιχεία τώρα για τα μεμονωμένα είδη βάσει των δεδομένων του 2011, της προηγούμενης χρονιάς. Από τα 4,5 εκατομμύρια λοιπόν βλέπετε με το μερίδιο των ζώων που μεταφέρεται για σφαγή, η πλειοψηφία μεταφέρεται βλέπετε για άλλους λόγους. Για τα ζώα τώρα που μεταφέρονται για σφαγή βλέπουμε ότι 500.000 το 11,54% αυτών ταξιδεύουν για λιγότερο από και περισσότερο από ταξιδεύουν 200.000, δηλαδή το 4,62% των ζώων που μεταφέρθηκαν το 2011, συγκεκριμένα. Τώρα, χείρι που έχουν μεταφερθεί για τη σφαγή εδώ έχουμε υψηλότερο αριθμό, αλλά και πάλι δεν φτάνει το 50%. Η μεγάλη πλειοψηφία των ζώων αυτών, γύρω στα 10 εκατομμύρια, 34% μεταφέρονται για λιγότερο των 8 ωρών. Πάνω από 8 ώρες, 2 εκατομμύρια ζώα, 6,8% του συνολικού αριθμού. Πρόβατα. Τα πρόβατα μεταφέρονται κατά κύριο λόγο για σφαγή. Βλέπετε το ροζ κομμάτι της πίτας που είναι μεγαλύτερο και το μερίδιο των ζώων τα οποία μεταφέρονται είτε για λιγότερο είτε για περισσότερο των 8 ώρων ε, είναι λίγο πολύ το ίδιο λίγο λιγότερο είναι το ποσοστό για τα ζώα που μεταφέρουν λιγότερο από 8 ώρες, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ζώα, συνολικός αριθμός ζώων που μεταφέρονται για σφαγή είναι πολύ μικρός, 120.000 είναι το συνολικό, το συνολικός αριθμός. Λιγότερα ε, είναι τα ποσοστά των ζώων που μεταφέρονται για ε, σφαγή, λιγότερο από 25%. Εδώ βλέπουμε ότι μεταφέρονται για περισσότερο από κυρίως γιατί, όπως φαντάζεστε, ο προορισμός τους είναι κυρίως η Ιταλία. Όπως σας είπα, υπάρχουν τεράστιες δοκιμάσεις και μεταξύ των ε, ειδών, αλλά και μεταξύ προέλευσης προορισμού. Βλέπετε ποιες είναι οι χώρες προέλευσης και οι χώρες προορισμού, οι σημαντικότερες. Κυρίως λοιπόν τα ζώα μεταφέρονται από Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία και Βέλγιο και μεταφέρονται προς Ισπανία, Ιταλία και κάτω χώρες. Και αυτό καλύπτει πάνω το 55% της συνολικής μεταφοράς ζώων. 2,5 εκατομμύρια κεφάλια. Για τους χείρους διαφέρει κατάσταση. Η μεγάλη πλειοψηφία, το 67% 20 εκατομμύρια χείρων, προέρχονται από τη Δανία ή από τις κάτω χώρες και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας είναι η Γερμανία που εισάγει το 5% περίπου του συνολικού ενωσιακού εμπορίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για τους χείρους. Παραλαμβάνω, ε, μάλλον σας ε, επισημαίνω ότι πρόκειται για το μέσο όρο για τα έτη 2005 έως 2009. Άλογα, κύριες χώρες προέλευσης Πολωνία, Γαλλία, Ρουμανία και Ισπανία, που καλύπτουν περίπου το 70% των εξαγωγών και εισαγωγής, όπως σας είπα, είναι κυρίως κατά κύριο λόγο Ιταλία με πάνω από το 50% και ακολουθεί με 30% των, ε, των ε, λόγων η Γαλλία. Εν συντομία λοιπόν ε, αυτά είναι τα στοιχεία, ελπίζω να είναι χρήσιμα για εσάς. Στοιχεία λοιπόν που αφορούν και του, το μέγεθος του εμπορίου αλλά και τα ποσά, τα ποσοστά, των ζώων που μεταφέρονται για διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο των οκτώ ωρών. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και φυσικά θα παρακολουθήσουμε και την όλη συζήτηση. Molto Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση και για την σαφή αυτή επισκόπηση που μας δώσατε για τα ευθυντικά στοιχεία αυτά. Και τώρα να δώσω τον λόγο στον Αντιπρόεδρο. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, zacznę od podziękowań. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και λάβαμε όλα τα στοιχεία αυτά που μπορούσαμε να λάβουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πληροφορίες πάρα πολύ σημαντικές, γιατί μας κάνουν να γνωρίζουμε πιο πολλά σε ό,τι αφορά την μεταφορά των ζώων. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ καλή παρουσίαση όλων αυτών των πληροφοριών. Από δική μου πλευράς, ως εισηγητής, θα σας πω ότι επιμένω σε αυτά που είχα δηλώσει και κατά το παρελθόν στη συζήτησή μας. και υπό το φως της παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξακολουθούν να ισχύουν αυτά που είχα προτείνει ο εισηγητής. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ζώων για σφαγή. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε ό,τι αφορά τον προορισμό τέτοιων μεταφορών. Τώρα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά ζώων για άλλους σκοπούς, πέρα από τη σφαγή, τα προβλήματα δεν είναι τόσο μεγάλα όσο στην περίπτωση των ζώων που μεταφέρονται για σφαγή. Νομίζω ότι η κλίμακα των μεγάλων αποστάσεων μεταφοράς δεν αποτελούν τόσο μεγάλο ζήτημα. Μεταφορές που διαρκούν 20 ώρες δεν αποτελούν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, οι μεταφορές που διαρκούν πιο πολύ από 8 ώρες αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη παρουσιάσει την χρωματοδότησή του και εγκρίναμε και μια γραπτή δήλωση πριν από κάποιο καιρό. Μου προκάλεσε κάποια έκπληξη αυτά που είπε ο Επίτροπος στην τελευταία συνάντησή μας όταν δήλωσε ότι θέλει να περιορίσει το πεδίο εφαρμογή τη σχετική προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν ε, μπορεί να περιοριστεί μόνο στην προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, γιατί εδώ ε, εμπλέκονται και άλλες πτυχές οικονομικής ε, φύσης. Αλλά ας μην επαναλάβω αυτά που έχω ήδη πει. Σας ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε Γιάννους για τις δηλώσεις αυτές και δύο συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επισκόπηση αυτή που μας έδωσε και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον θα μπορούσαμε να λάβουμε πιο ε, εις βάθος πληροφορίες για τα αριθμητικά αυτά στοιχεία. Θα ήθελα να ξέρω δηλαδή ανατύπω ζώου και ανακράτος μέλος. Τι, ποιοι είναι οι λόγοι μεταφοράς ε, σφαγή ή μη. Αυτό λοιπόν ζητώ από την ε, Επιτροπή, λέει η κυρία Ντελάνγκε. Δεύτερη Ντελάνε. δευτερη ερωτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ακολουθήσουμε την λογική του Επιτρόπου Νταλή, το είπε και ο προηγούμενος ομιλητής την προηγούμενη εβδομάδα. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν τη λογική αυτή, τα στοιχεία αυτά είναι τελείως ε, μη σχετικά. Γιατί η νομοθεσία λειτουργεί σωστά και το μόνο που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι οι όροι, οι συνθήκες μεταφοράς των ζώων και όχι ο λόγος μεταφοράς τους. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία που ακολουθεί ο κύριος Ντάλει. Θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Προφανώς μπορούμε να κρατήσουμε την τρέχουσα την νομοθεσία, στην οποία περίπτωση όμως θα πρέπει να βελτιώσουμε τον έλεγχο και την εφαρμογή της. Αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε, γιατί αν θέλουμε ένα σύστημα όπως αυτό που φαίνεται ότι θέλει ο κύριος Ντάλι, δηλαδή να κοιτάξουμε το θέμα των όρων, των συνθήκων μεταφοράς και όχι τόσο των όρων μεταφοράς, θα πρέπει να βελτιώσουμε τους όρους ε, εφαρμογής προκειμένου να αποφύγουμε την ε, κατάσταση που εμφανίζεται σε πολλέ περιπτώσει σήμερα, όπου για παράδειγμα κάποιε μεταφορέ αποφεύγουν την Αυστρία γιατί ξέρουν ότι είναι πιο αυστηρή η έλεγχη. Μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα εγγυηθεί, να μα υποσχεθεί ότι θα είναι πιο αυστηρό ο έλεγχο και η εφαρμογή τη νομοθεσία και πώ θα το εγγυηθεί αυτό, εφόσον είναι τα κρατημέλη υπεύθυνα και εμεί, πώ θα έπρεπε να αλλάξουμε σύστημα τελικά και να επιβάλλουμε παρόλα αυτά ένα χρονικό όριο. Κύριο Σμίτ και ο κύριο Κάπουλα Σάντο στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Ντελάνγκε. Ε, είναι λογική η διατύπωση και θα ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί πραγματικά είναι λεπτό το ζήτημα και συναισθηματικά φορτισμένο. Απηχώντα την παρέμβαση τη κυρία Ντελάνγκη, μα έχει δώσει κάποια στοιχεία περισσότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως το σημαντικό είναι γιατί μεταφέρω σε τόσο μεγάλες αποστάσεις ε, ε, τα ζώα. Ε, δεν έχουμε αρκετά σφαγεία σε, όλα, σε όλες τις περιοχές επειδή ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο. Εξηγήστε μας. Η δική μου πολιτική ομάδα δεν ομονοεί. Υπάρχει διάσταση απόψεων για αυτό το θέμα. Πάντως, ε, ο πυρήνας της έκθεσης είναι η παράγραφος 8 και λέει ο εισηγητής ξεκάθαρα ότι ο κανονισμός όσο έχει τώρα δεν έχει λειτουργήσει εύρυθμα και άρα θα πρέπει να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό και αν εφαρμόζεται σωστά σε όλα τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται αναθεώρηση και κυρίως θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα μικρά τοπικά σφαγεία, το ίδιο και για τις μονάδες επεξεργασίας ε, κρέατος, δηλαδή τα ε, σφαγεία να πηγαίνουν από τα, ε, τα σφάγια, συγγνώμη, πηγαίνουν από τα σφαγεία κατευθείαν στις μονάδες επεξεργασίας. Γι' αυτό σας μιλούσα για το οικονομικό μοντέλο. Δεν είναι βιώσιμη η μέθοδος που ακολουθείτε. Γι' αυτό και έχω καταθέσει διάφορες τροπολογίες γιατί ιδιαιτέρως για τον αριθμό ε, των ορών μεταφορές. Έχουμε από ε, τον Ιανουάριο του 2011 συστάσεις ε, του ΕΦΣΑ για τα άλογα συγκεκριμένα, για τους τάβλους κτλ. Ε, και άρα θα πρέπει πέρα από όλα τα προηγούμενα που σας είπα να εξετάσουμε και τις ε, κρατικές επιδοτήσεις ε, καθώς και τους υγειονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο στις μικρές μονάδες ε, τα συστήματα εξαερισμού, ε, να εφαρμόσουμε τι εκείρωσεις σε περίπτωση παραβίαση ε, των κανόνων του κανονισμού, όπω παραδείγματο χάρη στην έκθεση που κάναμε για την, το ευζήν των ζώων. Επίση, χρειάζεται καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένε φορέ. Τα υποχρεωτικά συστήματα με σαφή κυρώ μα βοηθούν να τηρούμε τα ορόσημα. Χρειαζόμαστε ούτω ή άλλως μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να γίνονται γίνονται σωστά οι έλεγχοι επί τόπου, ένα ξεκάθαρο διαφανή μηχανισμό εφαρμογή σε επίπεδο κράτου μέλου, αλλά γι' αυτό χρειάζομαστε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Επίση, ανταλλαγή βελτίζων πρακτικών, με ποιο τρόπο κάποιοι εφαρμόζουν σωστά με και άλλοι όχι. Επίση, ε, σεμινάρια, κατάρτιση, επιμόρφωση για τα ζητήματα αυτά. Ε, αυτά τα στοιχεία νομίζω θα διευκρινίσουν και θα ενισχύσουν το περιεχόμενο της έκθεσης. Πάντως θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγητή για τη διατηρεί την ισορροπία παρά ε, τη συναισθηματική φόρτωση αυτού του ζητήματος. Ευχαριστούμε. Λουίς Κάπουλα Σάντος και μετά Άγνιο παρακαλώ. Ευχαριστώ θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος ε, της πολιτικής μου ομάδας ε, και της κυρίας Κάρντενμπαχ που είναι η ισχυώδης εισηγήτρια της ομάδας μας. Δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα και μου ζήτησε να μεταφέρω τις παρατηρήσεις σα ε, πρώτον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλη τη δουλειά που έκανε και τον τρόπο με τον οποίο πρωτού συντάξει καν τη γνωμοδότηση συνεργάστηκε με όλους τους ενδιαφερομένους. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που η ομάδα μου θεωρεί σημαντικά και θα καταθέσουμε σχετικέ τροπολογίε. Ε, κάποια αναφέρθηκαν από τον συνάδελφο Σμίδε... αλλά θα ήθελα και εγώ παρόλα αυτά να τα σχολιάσω. Η κυρία Κάρντενμπαχ ανησυχεί όλο ιδιαίτερο για τον αριθμό των ζώων που μεταφέρονται από τη μία χώρα ε, στην άλλη, διότι στη χώρα προορισμού ε, μπορούν να λάβουν τη σήμανση προέλευσης. Αυτό ε, το στοιχείο δεν είναι τόσο γνωστό ε, και πιστεύω ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αναλυθούν για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Η κυρία Κάλενμπαχ επίσης συμφωνεί με τον εισηγητή για την ανάγκη να διατηρηθεί ένα δίκτυο μικρών ασφαγείων γιατί τα πρότυπα ασφάλειας ε, και οι υγειονομικές συνθήκες ε, ε, θα πρέπει να τηρούνται σε αυτές τις μικρές, μικρές μονάδες. Ε, και έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την ε, ε, μεταφορά των ζώων σε μεγάλες αποστάσεις για μεγάλο αριθμό ωρών είναι ισοσκελισμένη θέση του εισηγητή, όπω σα έλεγα στην αρχή τη παρέμβασή μου, αλλά σχετικά με τον αριθμό των ωρών Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα σε κάποιε εξαιρέσει που σχετίζονται με γεωγραφικά ε, χαρακτηριστικά χωρών, όπω η δικιά μου ε, είναι διασκορπισμένα τα κέντρα και γι' αυτό το λόγο ορισμένε φορές χρειάζεται μεταφορά για μεγαλύτερο αριθμό ωρών. Θα πρέπει λοιπόν κάποιε εξαιρεσει να ληφθούν εδώ υπόψη και ευχαριστώ τον εισηγητή που αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα ε, η διαθεσιμότητα των εναρμονισμένων δεδομένων είναι το επόμενο θέμα και η εναρμόνιση των υφιστάμενων κανόνων ε, εφόσον ε, όπως ήδη ακούσαμε υπάρχει μεγάλη διαφορά από κράτος σε κράτος ως προς την εφαρμογή του κανονισμού χρειαζόμαστε λοιπόν εναρμόνιση ως προς ε, τους κανόνες ε, εφαρμογής του κανονισμού και κλείνοντας να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή και να ε, υπενθυμίσω ότι θα θέσουμε διάφορες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και φυσικά θα συνδυαστούν με τροπολογίες άλλων συναδέλφων που ενδεχομένω να συμπαραταχθούν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε Λουίς άγνιο και μετά ο Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να επαναλάβουμε κάποια από τα στοιχεία τα οποία έχουμε πει και στο παρελθόν. Λάθος η προσέγγιση. Υπάρχει η αντίληψη ότι αν περάσει το Κοινοβούλιο τέτοια ε, νομοθεσία για τη μείωση ε, των, ε, του, της ώρας μεταφοράς, θα είναι αρνητικές οι επιπτώσεις. Να σας πω το εξής για έναν εκτροφέα που έχασε ένα ζώο θεώρησε ότι το έχασε και μετά από μήνες το βρήκε μεταξύ όρθιο σε παγιδευμένο σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να ξεφύγει. Ωστόσο, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες για τα ζώα αυτά όταν μεταφέρονταν γιατί τα αναγκάζουν σε μυρικασμό και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Άρα, το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ανάμιξη των ζώων αυτών και υπερβολικός μεγάλος πληθυσμός των ζώων κατά τη μεταφορά αποτελούν τα βασικά προβλήματα και δεν χρειάζεται καν να σταματήσουμε τα φορτηγά για να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Οι ελεγκτές και οι επιθεωρητές μπορούν να το διαπιστώσουν και κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση. Έχουμε στο Ενωμένο Βασίλειο τα, μια σχετική υπηρεσία για την καταγραφή και την εποπτεία της ευημερίας των ζώων. Και είναι μεγάλη τροπή για κάθε Βρετανό να μην πλήρει τέτοιους όρους των σχετικών υπηρεσιών. Ένας ε, εκτροφέας ε, μάλιστα αυτοκτόνησε όταν αποκαλύφθηκε ότι ένας από τους υπαλλήλου του κακό μεταχείριζε όταν είναι ζώο. Αυτό το θέμα κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει στην Ολομέλεια όπου ψηφίζουν 45 ε, ευρωβουλευτές. Στην Ισπανία βέβαια ανέχονται και τις σταυρομαχίες για λόγους διασκέδαση. Εγώ δεν θέλω εκπρόσωποι της χώρας αυτής ε, να κάνουν νομοθεσία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θέλουμε άλλους νόμους, θέλουμε καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων. Η κυρία Πάουλσεν, ε, η αντιπρόεδρος μας. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας. Είναι εξαιρετική η έκθεση του, ιδιαίτερα ε, ίσως και Νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε διάφορα επιμέρους ζητήματα και όχι μόνο σε αυτό το 8ωρο της μεταφόρας. Ε, πιστεύω ότι παρά είναι τετράγωνος ο τρόπος ε, που ε, ε, προσεγγίζουμε το θέμα και δεν αποκαλύπτουμε ολόκληρη την αλήθεια. Χρειαζόμαστε αυστηροποίηση των κανόνων και καλύτερη τήρηση των κανόνων. Σε αυτό έγκυται η αδυναμία και οι ελλείψεις μας. Το τελευταίο σκάνδαλο που έγινε με τη μεταφορά ε, των ζώων ε, από την Ανατολική Ευρώπη προς την Τουρκία όπου τέσσερις ε, σοβαρότετες οργανώσεις προστασίας των ζώων καταδίκασαν την μεταφορά. λοιπόν, κατά δύο τρίτα, παρότι παρακολουθούσαν αυτή την μεταφορά αυτές οι οργανώσεις, κατά δύο τρίτα δεν εφαρμόστηκε το κεκτημένο, οι κανόνες που αυτή τη στιγμή ισχύουν. Οπότε... Καταλαβαίνουμε ότι ε, το 30% λειτουργήσε. Ε, λοιπόν, σε σχέση με το παρελθόν είναι φοβερή πρόοδος. Έτσι μας λένε. Τι σημαίνουν όλα αυτά ότι παρόλα αυτά που ακούγονται έχουν νόημα αυτά που κάνουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, προσπαθίες μας για να ανέβουμε αυτό το 30% και να τίνουμε προς το 100% και θα πω ότι ε, η λέξη κλειδί είναι εφαρμογή, εφαρμογή και εφαρμογή, καλή τήρηση των κανόνων γενικότερα και όχι μόνο σε σχέση με το 8ωρο υπάρχουν αρκετά δυνατοί υπολογιστές, ε, υπολογιστές συγγνώμη, πλέον που θα μπορούσαν να ελέγχουν ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις μεταφορές ε, των ζώων. Αναρωτιούνται κάποιοι γιατί παίρνει τόση ώρα η μεταφορά ανάμεσα ε, στα σφαγεία. Στα περισσότερα κράτη-μέλη μειώνεται δραστικά ο αριθμός ε, των μικρών σφαγείων. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτή η ε, εξέλιξη περιορίζει αλλά με ε, ριζικό τρόπο την δυνατότητα επιλογής των εκτροφέων. Σε πολλές περιοχές έχουν μόνο ένα σφαγείο στο οποίο μπορούν να μεταφέρουν τα ζώα τους και καταλαβαίνετε ότι αυτό πλήττει την ανταγωνιστικότητα νομιμότητα αυτών των ε, εκτροφέων γιατί δεν έχουν επιλογή. Όταν μιλάμε τώρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου και εν ώψη της μεταρρύθμισης κοινής γεωργικής πολιτικής ε, θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να καταβάλουμε μεν προσπάθειες να διορθώσουμε την κατάσταση αλλά όλα αυτά τα μέτρα που σχετίζονται με τη διατήρηση των μικρών σφαγιών μου δημιουργούν διασμούς. Καλύτερα θα ήταν να διερευνήσουμε ε, τις, ε, τα αίτια, για ποιο λόγο ε, εξαφανίζονται αυτά τα μικρά σφαγεία, με ποιο τρόπο μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα διευκολύνοντας την λειτουργία αυτών των σφαγείων και ευνοώντας έτσι και τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των εκτροφέων στην Ήπεθρο. Ε, για τους υγειονομικούς ε, κανόνες, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό το 8ωρο. Ε, το πρόβλημα με τους υγειονομικούς κανόνες είναι θέμα επιληρωμής, ε, διότι οι υγειονομικοί κανόνες σχετίζονται με τους ε, ελέγχους. Είναι υπερβολικά υψηλό το τέλος που αντιστοιχεί στον έλεγχο ανακυλό ε, κρέαντος. Και άρα είναι επαχθέστατο το τέλος αυτό για, τους, για τα μικρά σφαγεία και άρα εξαφανίζονται. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά επιμέρους ζητήματα. Θα ήθελα ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή γιατί κατέβαλε σοβαρότατες προσπάθειες ε, να βρει μια ισορροπία για αυτό το τόσο δύσκολο θέμα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστούμε ε, κυρία Πάουλσεν. Ε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς, ε, κυρία Ράιμερς, να πω ότι το θέμα δεν είναι μόνο η ώρα της μεταφοράς, ε, η μεταφορά των ζώων για σφαγή ε, μάλλον η μεταφορά γίνεται όχι μόνο για σφαγή, αλλά και για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα διάμεση σταθμή, επειδή δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εκτροφές σε ένα εκτροφείο. Άρα είναι πάρα πολύ γενικό το να ορίσουμε ένα όριο 8 ωρών. Γιατί αν είμαστε τόσο απόλυτοι ε, σε αυτό το τομέα, μπορούμε να είμαστε τόσο απόλυτοι και σε άλλους τομείς. Δεν το κάνουμε αυτό παντού. Η εκτροφή, η μορφή των εκτροφίων είναι διαφορετικό, διαφορετική. Και έχουμε χώρες με μεγάλα, μικρά εκτροφία και όλα αυτά έχουν σημασία. Βλέπουμε για παράδειγμα στους κύριου και στα πουλερικά η ώρα μεταφοράς είναι σε υψηλό ποσοστό κάτω από 8 ώρες. Αυτό έχει να κάνει ότι έχουμε εκτροφία με μεγάλους πληθυσμούς. Δεν συζητάμε εδώ στο σημείο ότι η ώρα μεταφοράς ξεκινάει από τη στιγμή που φορτώνεται το πρώτο ζώο. Θα θυμάστε ότι για τα πρόβατα, για παράδειγμα, ε, για να φορτώσει κανείς ένα φορτηγό γεμάτο με πρόβατα, πρέπει να περάσει σε διάφο από διάφορα εκτροφία. Άρα έχουμε και τον όρο και τον χρόνο φόρτωσης, ο οποίος παίζει μια σημασία. Τι γίνεται με τις περιοχές όπου υπάρχουν πάρα πολύ μικρά ε, διασκορπισμένα εκτροφία αυτές τις περιπτώσεις ε, ε, αν ορίσουμε έναν μέγιστο χρόνο φόρτωσης και μεταφοράς, ε, θα υποστούν αρνητική διάκριση, γιατί θα εκτοξευτούν στα ύψη το, τα έξοδα. Αν υπάρχει, για παράδειγμα, και μεγαλύτερος κίνδυνος μόλυνσης. Μήπως ε, λοιπόν δεν είναι υπεύθυνο ο τρόπος αυτός δράσης και μήπως θα πρέπει να εστιαστούμε πιο πολύ στους όρους και στις συνθήκες μεταφοράς, όπως και στους ανθρώπους για παράδειγμα. Ε, άλλο να ταξιδεύουμε με ένα καλό και υψηλή ποιότητα τρένο και άλλο να ταξιδεύουμε υπό άλλες συνθήκες. Είναι λίγο υπερβολικά απλοϊκός ο τρόπος υπολογισμού μόνο με τις ώρες μεταφοράς. Και θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε τι γίνεται για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν, για παράδειγμα, οι εκτροφή στην επιλογή ε, σφαγείων. Όταν υπάρχει, για παράδειγμα, προβλήματα στην εφαρμογή νομοθεσίας ή προβλήματα με τους υπαλλήλους, γιατί, για παράδειγμα, τα μικρά εκτροφία χρειάζονται ε, εξειδίκευση σε εργατικό δυναμικό το οποίο δεν είναι πάντα εξίσου εύκολο. Αυτό παρουσιάζει λοιπόν τεράστια προβλήματα και εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε να υπάρχει πρόσβαση και για τον εκτροφέα στην αγορά γιατί αν ορίζονται όλα αυτά υπερβολικά δεν υπάρχει περιθώριο δράσης ως επιχειρηματίας πλέον γιατί θέλουμε αγρότες οι οποίοι θα έχουν μια συμπεριφορά επιχειρηματία αυτό το λέμε πάντα. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ως ε, παράγοντα. Να προσέξουμε λοιπόν τελικά μην καταλήξουμε να συγκρίνουμε ανώμια σχήματα. Τι γίνεται με τις ε, ελεύθερες μεταφορές ζώων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται αλλά και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθεί και με τις ομάδες πίεσης, να δούμε τι γίνεται, δηλαδή όχι μόνο στο γεωργικό κλάδο, αλλά και στον, ε, στους υπόλοιπους κλάδους. Θα συζητήσουμε λοιπόν εκτεταμένα την έκθεση αυτή και θα βρούμε έναν τρόπο, φαντάζομαι. Φαίνεται ότι όλοι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εστιαστούμε κυρίως σε θέματα ποιότητας και στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, γιατί είναι γεγονός και πρόβλημα άλλωστε ότι όλο και πιο πολλά κοινά υπάρχουν στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ, Μπρίτα Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω όλα τα επιχειρήματα για την εφαρμογή. Τα έχουν πει και προλαλήσαντε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξέρω ότι η Κομισιόν και ο Επιτρόπος ήρθε εδώ ε, έδειξε ότι πλέον απελπίζεται όταν τον για κάτι που δεν μπορεί να κάνει. Μα το θέμα επανέρχεται συνεχώς διότι τελικά δεν επιτυγχάνεται τίποτε. Οπότε δεν θα ήταν πια ένα αγκάθι στο πλευρό του το θέμα, αν έκαναν κάτι τελικά γι' αυτό. Έχω υπόψη να καταθέσω τροπολογίες που έχουν να κάνουν πιο πολύ με τον περιορισμό ε, του χρόνου μεταφοράς ε, των ζώων και ιδίως ε, των ε, υποειδών. Θα έλεγα, εάν εξεταστούν τα στοιχεία και η ΕΦΣΑ έχει εξετάσει τα στοιχεία αναλυτικά. Για το 2010 μία μελέτη Γκραντά, Μόρλιν 11 και άλλες ε, μελέτες αναρρυθμητές που δείχνουν ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ συγκεκριμένα και με διαφορετικό τρόπο το ζήτημα της μεταφοράς ε, των υποειδών και όχι όπως αντιμετωπίζεται τη μεταφορά άλλων ζώων. Είναι καιρός πλέον να πάρει η Κομισιόν τα απαραίτητα μέτρα για τη μεταφορά των ε, αλόγων που μεταφέρονται για σφαγή. Όταν μεταφέρονται για άλλους λόγους, επειδή είναι ένα ακριβό ζώο, ε, δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί, ε, τα προσέχουν ιδιαίτερα. Αλλά είναι σκάνδαλο η μεταφορά των αλόγων όταν πηγαίνουν για σφαγή. Ξέρουμε ότι μπαίνουν από τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης, από την Ουκρανία, τη Ρωσία, μπαίνουν ε, στις διάφορες χώρες, φορτώνονται σε φορτηγά και πηγαίνουν στη Σικελία όπου σφαγιάζονται. Δεν πρέπει να το ανεχτούμε αυτό, πολύ απλά. Και ο πιο απλός τρόπος ε, είναι να έχουμε κάποιες ε, διατάξεις για τη μεταφορά όταν κάποιος περνά και βλέπει τα ζώα αυτά στην Ιταλία να σκεφτεί λίγο τι έχουν περάσει για να φτάσουν εκεί. είναι μέτρα που πρέπει να ληφθούν και δεν επηρεάζουν τη γεωργία σε μακρά κλίμα, μεγάλη κλίμακα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Επιτροπή είναι ενωμένη το ότι θέλει υψηλά πρότυπα ε, για τη μεταφορά των ε, ζώντων ζώων. Αλλά ο περιορισμός του χρόνου μεταφοράς 8 ώρες ανά ταξίδι είναι κατά την άποψή μου ένα αμβλή ε, εργαλείο. Δηλαδή δεν θα πετύχει κατά ανάγκη τους στόχους αυτούς για την καλή μεταχείριση και την ε, ευζοία των ζώων. Αν είναι κακές οι συνδίκες μεταφοράς, ε, οδικής μεταφοράς των ζώων, τότε και μια ώρα είναι πολύ, πολύ χρόνος. Αλλά εάν οι, όροι, οι μεταφοράς είναι ποιοτικέ, είναι ικανοποιητικέ, στηρούν κάποια ικανοποιητικά πρότυπα, αν τα ζώα για 10 ώρες ε, ταξιδεύουν, αλλά με τέτοιες συνθήκες, αυτό δεν είναι αγχογόνο. Είναι πολύ λιγότερο από ότι να κάνουν ένα ταξίδι 8 ε, ωρών όπου τα ανεβάζουν, τα κατεβάζουν ε, και μετά τα ξαναφορτώνουν σε ένα άλλο φορτηγό για άλλες δύο ώρες. Παναλαμβάνω μπορεί να χάσει την αποτελεσματικότητά του το μέτρο αν δεν το εφαρμόσουμε σωστά. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε και την ανάγκη, ε, το λόγο που γίνονται πολλά ταξίδια. Έχω εμπειρία προσωπικά και λόγω της δικής μου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εξασφάλιση ποιοτικών προτύπων, κάτι που απαιτούν οι μεγάλοι λιανοπολιτές, ε, σημαίνει ότι ουσιαστικά θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο επί των σφαγίων και γι' αυτό πολλές φορές απαιτούν ε, τη μεταφορά των ναζών για πολλές ώρες γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιείται ένα-δύο το πολύ εγκεκριμένα σφαγεία ε, για τα προϊόντα ε, των λιανοπολιτών. Η ζήτηση, μάλλον το, να ζητήσουμε να υπάρχουν τοπικά μικρά σφαγεία νομίζω ότι ούτε οικονομικό είναι ούτε θα έχει κάποια μεγάλη επίπτωση. Αλλά νομίζω συμφωνούμε όλοι, δεν χρειαζόμαστε περισσότερου κανόνε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει οικουμενική εφαρμογή αυτών των κανόνων και στα 27 κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο κύριο Βοητσιακόφσκι για την έκθεσή του. Και πράγματι θα πρέπει, όπω είπε και η Κομισιόν και πολλοί συνάδελφοι, να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των ζώων που μεταφέρονται για σφαγή και των ζώων ε, που μεταφέρονται προ άλλα ε, αγροκτήματα, προ πάχυνση ή τέλο πάντων για να συνεχίσουν τον κύκλο ζωή του με άλλο τρόπο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε, κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στο σημείο 9 γίνεται η διάκριση. Δηλαδή μιλάμε για το χρονικό των οκτώρων για τη μεταφορά ζών προς φαγή. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας αγαπητοί συνάδελφοι. Άκουσα με πολύ προσοχή τα σχόλιά σας, τα περιμένω να δω και τις τροπολογίες σας. Νομίζω ότι όλοι στο ίδιο μήκο κύματο ε, βρισκόμαστε και νομίζω ότι με κοινέ προσπάθειες ε, θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε μια καλή γνωμοδότηση. Θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε ένα πρόβλημα, το οποίο έθεσαν αρκετοί συνάδελφοι. Ίσως ο κύριος Σμίθ ήταν ο πλέον ξεκάθαρος. Δεν μιλάμε μόνο για τη μεταφορά. Υπάρχει και ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο. Αλλά και γενικότερα ίσως οι συνδικές μεταφορέ επηρεάσουν αυτό το οικονομικό μοντέλο σε κατεύθυνση που να είναι πιο ε, θετική για την ε, γεωργία και την κτηνοτροφία. Δεν θέλουμε να υπάρχει συγκέντρωση σε τεράστια εργοστάσια μεταποίησης ε, και επεξεργασίας όπου τα ζώα φτάνουν έχοντας διανύσει τεράστιες αποστάσεις. και βλέπουμε να εξαφανίζονται τα μικρά σφαγεία που πλήν ανταγωνιστικά ήταν σημαντικά για τους ε, κτηνοτρόφους. Το θέμα είναι να υπάρχει επιλογή, να μην υπαγορεύεται ε, στον κτηνοτρόφο το που θα πουλήσει τα ζώα του. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω κάτι, αν είναι δυνατόν. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να δούμε τον αριθμό των εταιριών των μικρών σφαγείων. Πόσα τέτοια μικρά σφαγεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και πώς έχει μεταβληθεί η κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες. Τέτοια στοιχεία θα μπορούσαν να είναι πολύ ενδιαφέροντα στη δική μου χώρα την Πολωνία αυτή η διαδικασία, ότι δηλαδή εξαφανίζονται σιγά σιγά τα τοπικά σφαγεία, ε, παίρνει πολύ γρήγορες, ε, μάλλον παίρνει πολύ γρήγορου ρυθμού. πάρα πολύ γρήγορα εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο. Και αυτό δεν ήταν, ε, επειδή δεν μπορούσαν να τηρήσουν ε, τα πρότυπα, αυτό δεν ήταν ευεργετικό για τον γεωρικό και εκτροφικό τομέα της χώρας μου. Πριν λοιπόν λάβουμε μια τελική απόφαση, και πριν εξετάσουμε και τις τροπολογίες, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει τα σχετικά στοιχεία για να δούμε πώς έχει αλλάξει η κατάσταση, πόσα σφαγή έχουμε τώρα, ε, πόσα είχαμε πριν. Τις τελευταίες δεκαετίες, να δούμε πώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι μέχρι τις 30 Μαΐου 12 το μεσημέρι μπορούν να καταθέσουν στις τροπολογίες τους. Περνούμε τώρα στην, στο επόμενο σημείο. Η Επιτροπή θέλει το λόγο. Η κυρία Ντελάουν σα είχε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Αν δεν θέλετε. Καλά. Θα το δείτε διμερός. Ε, σημείο 4, κοινή οργάνωση αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα, ενιαία ακόα. Πρόκειται για την τρίτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Ίσως δεν έχουμε δώσει τη δέουσα σημασία σε αυτό το σημείο της ε, μεταρρυθμιση κοινή γεωργικής πολιτικής. Καλό θα ήταν ο κύριος ε, Νταντά να μας υπενθυμίσει τις βασικές του ιδέες. Θα δώσω το λόγο στον ε, Μισελ για να αρχίσει η συζήτηση έτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση για την ΚΟΑ και θα πω ακριβώς αυτό που πιστεύω φαίνεται να μην ε, ενδιέφερε κανέναν μέχρι πριν από λίγες μέρες ε, όπου το βρίσκουν όλο αυτό το ζήτημα συναρπαστικό και παθιάζονται κιόλας. Παρ' όλα αυτά είναι αμπηγός νομικό το κείμενο. Ως εκ τούτου χρειάστηκε πολλή δουλειά για τα νομικά ζητήματα θα βοηθήσω λοιπόν τους συνεργάτες μου, παρεπιπτόντως ε, τον, ε, τους βοηθούς μου και την Ελένα από τη γραμματεία ε, της Επιτροπής. Να προσπαθήσω να πω τα πράγματα απλά. Προτείνω μέσα στην έκθεσή μου να επανεισαγάγουμε τρία ζητήματα, τρεις φακέλους που ε, εσχάτως έχουν εγκριθεί ε, μεταξύ άλλων και στους τριμερείς διαλόγους ε, το πακέτο γάλακτος. Θέλω να επανέλθει στην κοινή ΚΟΑ. Επίσης, η συνάδελφος Γκαρσία Περέζα ασχολείται με το θέμα των κανόνων θέσης σε εμπορία. Θέλω και αυτό το ζήτημα να επανενταχθεί μέσα στην ΚΟΑ μέσα στην έκθεση για την ΚΟΑ μάλλον. Και το τρίτο θέμα που τώρα εξετάζεται υπό την ε, ηγεσία του συναδέλφου Ντόρφμαν στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Αυτά τα τρία ζητήματα ε, αποτέλεσαν αντικείμενα εκθέσεων στην Επιτροπή μας. Έχει γίνει ψηφοφορία. Καλό θα ήταν Εφόσον έχουμε αποφανθεί για κάθε ένα, κάθε μία από αυτές τις ε, προτάσεις ε, ξεχωριστά, να περιοριστούμε ως προς τροπολογίες, ε, χωρίς βέβαια να απολέσουμε το βασικό δικαίωμα κάθε βουλευτή, δηλαδή να καταθέτει τροπολογίες για να επηρεάσει τις εξελίξεις. Παρότι κάποιοι θέλουν να επανέλθουν στα παρελθόντα, δεν προκύπτει πλειοψηφία για να επανέλθουμε στον τρόπο πλαισίωσης και παρέμβασης, ε, βαριάς δημόσιας παρέμβασης όπως στις δεκαετίες 70 και 80 στην αγορά ως εκ τούτου. Σημειώστε συνάδελφοι ότι μεταφέρουμε στους γεωργούς και στους τομείς ε, την ευθύνη να αυτοοργανωθούν και να διαχειριστούν τις ε, αγορές. Ανακολουθήσετε αυτό τον τρόπο ανάλυσης μέσα στην έκθεση. Θα έπρεπε να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών του κλάδου και να διευκρινίσουμε επίσης ε, τα θέματα του δικαίου του ανταγωνισμού. Προτείνω εφαρμογή του άρθρου 42 της Συνθήκης της Λισαβόνας που μας επιτρέπει μέσα από κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να αποκλίνουμε σε σχέση με το άρθρο 101 εδάφιο 1 ως προς το δίκαιο του ανταγωνισμού για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που μάλιστα περιγράφονται μέσα στην έκθεση οι γεωργοί λοιπόν και ο ίδιος ο κλάδος θα έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το τι είναι εφικτό, διότι σήμερα αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες οι οποίες ε, όμως αν κράτο, ε, την πολύ πολύ διαφορετικής μεταχείρισης από τις αρχές αρμόδιες για τον ανταγωνισμό. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε πέραν κάθε Σε Το εθνικό δίκαιο διαφέρει, είναι προφανέ ε, από κράτο σε κράτος ε, και άρα αρμόζει στο επίπεδο οργανώσεων, παραγωγών, διεπαγγελματικών οργανώσεων και δίκαιων δικαίου του ανταγωνισμού, ένα, ε, ε, μια μορφή εναρμόνισης. Ε, η γερμανική νομολογία, θα έλεγα μάλιστα το γερμανικό σύνταγμα, απαγορεύει την σύσταση διεπαγγελματικών ενώσεων όπως αυτές που βρίσκουμε στην Ιταλία λόγω της νομοθεσίας κατά των τραστ Πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος και άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξετάσουμε ε, τις ε, οικίες εθνικές διατάξεις ε, για όλα αυτά τα ζήτημα. Θα επανέλθω τώρα στα αυτά τα τρία ζητήματα επί των οποίων έχει απομφανθεί με σαφήνεια το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων και στην έκθεση του Αλμπερντές πέρυσι. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για το θέμα της ζάχαρης. Προτείνω να επανεισάγουμε το σύστημα των ποσοστώσεων μέχρι το 2020, ενσωματώνοντας και έναν επιπρόσθετο μηχανισμό, χάρη στον οποίο και ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά θα μπορούμε ε, να ε, ε, εισάγουμε ζάχαρη, που ε, υπέρ της ποσόστοσης ε, και ε, να περιορίζουμε αντίστοιχα την τροφοδοσία σε ζάχαρη κάτω από την ποσόστοση ανάλογα με τις ανάγκες. Υπάρχουν κάποιοι που αποδίδουν τα εύσημα χωρίς καν να έχουν διαβάσει την έκθεση μου. Θα ήθελα να σας μιλήσω συγκεκριμένα για την ημερομηνία 2020 και τα δικαιώματα φύτευσης. Προτείνω να επανέλθει λοιπόν το κείμενο με συγκεκριμένη ημερομηνία αντίθετα με αυτά που έλεγα στην αρχή, διότι ε, υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε προηγούμενη απόφαση δέχτηκε την παραβίαση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων διότι υπήρχε ε, ε, καταληκτική ε, πρόθεσμια για το μηχανισμό. Εγώ θα προτείνω 2030 και δέχομαι και πολύ πιο απομακρυσμένες ημερομηνίες αν το ζητήσουν κάποιοι άλλοι. Έχοντα συζητήσει με πάρα πολλού συναδέλφου. δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω αυτά που ήδη ξέρετε, θα σας πω μόνο ότι με την επανένταξη αυτού του τμήματο ανοίγει ο δρόμος για τις συμβαστικέ τροπολογίες, ούτω ώστε να αποτυπωθούν και τα πορίσματα τη ομάδα υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο μέτρο που αυτά και λυπούμε πάρα πολύ ε, να πω παρόδο ότι δεν συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, η Επιτροπή μας συμμετέχει, αλλά οι ίδιοι βουλευτές δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και λυπάμαι για αυτό. Σε σχέση με το γάλα, ε, δεν θεωρώ ότι ε, θα προσφέρουμε τελική λύση για την σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων και πάλι τώρα σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν από λίγες εβδομάδες θα ήθελα να σημειώσω το εξή. Αυτό το σύστημα που εγκρίναμε πριν από λίγες εβδομάδες λοιπόν θα αρχίσει να ισχύει 1η Σεπτεμβρίου του 2012 άρα δεν καταλαβαίνω αυτά τα σχόλια που διαπιστώνουν ε, μη ικανοποιητική λειτουργία του σύστηματος. Αντίθετα χρειαζόμαστε ένα τρόπο ώστε να θεσπίσουμε ένα μηχανισμό που θα ευνοεί τους γεωργούς ε, που ε, ε, σε θελοντική βάση μειώνουν την παραγωγή και αντίθετα οι μεγάλοι γεωργοί που προσπαθούν μεσούς της κρίσης να αυξήσουν την παραγωγή τους εκμεταλλευόμενοι τα περιθώρια κέρδους βρίσκονται τελικά σε καλύτερη ε, καλύτερη θέση σε σχέση με τους μικρούς γεωργούς. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας. Να ευχαριστήσω και τους κοιόδης, ε, διότι ε, είχαμε πολλές κατηδίαν συσκέψεις και δύο ομαδικές συναντήσεις μέχρι τούδε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Μισελ, λέει ο Πρόεδρος. Θα αρχίσουμε ευθύ αμέσω τη συζήτηση και η Ράς μπερέσκη στη συνέχεια Ταραμπέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Δαντάν για τη δουλειά του και για την ε, μέθοδο που ακολούθησε τις τελευταίες εβδομάδες σε ό,τι αφορά τους υπεύθυνους και τις συνομιλίες για την επιτεύξη μιας συνένεσης. Εν γέννη, συμφωνώ με τις απόψεις του σε ό,τι αφορά τα διάφορα θέματα, σε ό,τι αφορά το πακέτο για την ποιότητα. Θα ήθελα να ζητήσω να διατεθούν στην Επιτροπή μας πιο πολλές πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα αυτό. Βρισκόμαστε σε φάση συζήτησης ε, με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τα διάφορα συστήματα ποιότητα, σε ό,τι αφορά όμως τις, τα πρότυπα και την μετοπίζει θα πρέπει να επιτευχθεί μια συμφωνία. Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις μεταρρυθμίσεις ε, της ε, ΚΟΑ. ζητείται και από τις δύο εκθέσεις ουσιαστικά και τα πρότυπα εμπορίας ε, να είναι ε, τα κατάλληλα και να ενσωματωθούν ε, στο πλαίσιο της ΚΟΑ. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες ε, ανταγωνισμού, νομίζω ότι στη γενική συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής υπάρχει μια γενική συμφωνία των παραγωγών, ιδίω ε, σε ό,τι αφορά το ότι βέβαια ό,τι έχει να κάνει με τις άμεσες ενισχύσεις και την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι πολύ σημαντικό και εγγυάται το μέλλον του κλάδου και του τομέα. Αν όμω δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε και να δρομολογήσουμε τα μέσα εκείνα που θα εγγυώνται τις δίκαιες σωστέ τιμέ και θα αντιμετωπίζουν τις διακοιμάσει των τιμών των γεωργικών προϊόντων, πώς μπορούμε να αγγίθουμε το μέλλον του κλάδου και του γεωργικού τομέα. Όλα αυτά τα μέσα, τα εργαλεία, τα πρότυπα και τους κανόνες που μπορούμε να εντάξουμε στο πλαίσιο της νέας ΚΟΑ, όταν θα ορίζουμε και ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων και θα δίνουμε τη δυνατότητα ενίσχυσης του ρόλου των νόσων παραγωγών, άρα του διαπραγματευτικού ρόλου των ίδιων των παραγωγών ε, στην αλυσίδα αυτή αξία. αυτό είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τις οποίες ε, έχουμε αναφέρει. Και υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, θα δώσουμε πολύ πιο συγκεκριμένες ιδέες για τα εργαλεία και μέσα αυτά και θα φροντίσουμε να μην υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες των κανόνων ε, μεταξύ των κρατών μελών σε κοινωνικό επίπεδο. Τέλος, να πω ότι συμφωνώ με τις σκέψεις και την πρόταση του κυρίου Ντάντα για τη ζάχαρη ε, και για τα δικαιώματα φύτευσης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή τη διαδικασία προσαρμογής στην ανταγωνιστικότητα που για τους δύο τομές αυτούς να την εγγυηθούμε, να την βοηθήσουμε έχουμε τις ποσοστώσεις για τη ζάχαρη μέχρι το 2020. Αν καταφέρουμε να διατηρήσουμε τα δικαιώματα φύτευσης ε, και στους αμπελώνες, νομίζω θα είναι κάτι θετικό επίσης. Συμφωνούμε με τις ε, απόψεις του κ. Νταντάν και θα συγκεκριμενοποιήσουμε τις προτάσεις μας με τροπολογίες συγκεκριμένες ε, στην όλη διάρκεια της εξέτασης αυτής της έκθεσης. Πρέπει να απαντήσουμε, να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Στο θέμα της, ε, του πακέτου ποιότητας, νομίζω ότι καλή ιδέα είναι να μείνει ξεχαριστό κεφάλαιο το θέμα της, των ε, μεθοδών ποιότητας σε ό,τι αφορά τα πρότυπα εμπορευματοποίησης. Καλό θα ήταν λοιπόν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να κοιτάξουν το πρώτο τμήμα αυτό και ελπίζουμε το Συμβούλιο θα πάρει σχετική εντολή προς διαπραγμάτευση και προφανώς αν αυτό δεν συμβεί θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε αυτά τα σημαντικά στοιχεία τα ραμπέλα και μετά Ευχαριστώ πολύ. Έχω εργαστεί με τον ε, κύριο Νταντάν και ε, στο θέμα του γάλακτος και γι' αυτό μπορώ να συμφωνήσω με την αρχή που μας περιέγραψε, δηλαδή να έχουμε, μεγαλύτερη, να έχουμε μεταφορά περισσότερων εξουσιών ε, στον κλάδο. Θα επανέλθω να ενισχύσουμε λοιπόν την εξουσία των παραγωγών. Ε, πράγματι είναι σωστό και πολύ ουσιώδες. Δεύτερη μεγάλη αρχή, το άρθρο 42 της συνθήκης της Λισαβόνας ε, ε, δημιουργούσε παρέκκληση για τον ανταγωνισμό, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι, όπως είδαμε και με το γάλα, μετά την ψηφοφορία και τη συναπόφαση με το Συμβούλιο, είδαμε ότι οι πρώτοι που προσπαθούν να φρενάρουν το σύστημα που δύσκολα καταφέραμε να εφαρμόσουμε είναι η μεταπητική βιομηχανία. Όχι εξ ολοκλήρου, αλλά οι πιο πολλοί ε, προσπαθούν να πείσουν τους παραγωγούς να μην μπουν στο νέο σύστημα. Και όσοι δεν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι είναι αυτοί που ίσως ε, κινδυνεύουν περισσότερο. Θα πρέπει να Ξέρουμε ότι κάποιοι θα μας κατηγορήσουν για γραφειοκρατία, αλλά οι δημόσιες αρχές είναι αυτές που θα μπορούσαν ε, να είναι, αν θέλετε, αστιφυλάκα των αγορών. Και καλό είναι να υπάρξει μια ισορροπία για τη ζάχαρη και το γάλα. Τώρα, για τη ζάχαρη ε, χαίρομαι που άκουσα από τον ε, κύριο Νταντά να λέει ότι πρέπει να διατηρηθεί το σύστημα των ποσοστώσεων με κάποια βέβαια ελαστικότητα μέχρι το 2020. Καλό είναι αυτό. Για το 2030 για το κρασί τέλεια, το ίδιο. Τώρα όταν προτείνουμε το 2099, εντάξει δεν θα ζει κανένας από όλους είμαστε εδώ, αλλά τέλος πάντων τότε θα έχει αλλάξει το σύστημα. Για το γάλα μίλησα. Είδαμε την επικαιρότητα, τι έγινε μετά την ψηφοφορία. Υπάρχουν ε, πολλοί που έχουν ε, πιέσει ή παροτρύνει τους ε, παραγωγούς να μην μπουν σε αυτό το σύστημα. Προσοχή λοιπόν σε όλους τους τομείς παραγωγής υπάρχουν τα μεγάλα ολιγοπόλια ε, του τομέα της μεταπής βασικής παραγωγής και το πρόβλημα θα περάσει και σε άλλες παραγωγές σίγουρα. Οπότε θα πρέπει αρχές να είναι πολύ προσεκτικές ώστε να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες που από κοινού θα θεσπίσουμε. Grazie Mark. Albert poi Giovanni Lavia. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μισελ Τεντάν εξ ονόματος ε, του ΕΛΚ για το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Έχει απόλυτο δίκιο. Από νομικής άποψης είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα, το οποίο καλούμαστε να επεξεργαστούμε και νομίζω ότι η μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων συμφωνεί μαζί μου ότι μια γεωργία, ένα γεωργικό σύστημα ε, δεν, ε, ότι δεν, δεν ε, λειτουργεί το γεωργικό σύστημα, έχει αποτύχει. Αλλά πιστεύω ότι η εντελώς ελεύθερη διαμόρφωση του κλάδου και αυτή δεν θα λειτουργήσει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε στο μέλλον μια κοινή οργάνωση αγορά. Και γι' αυτό λοιπόν τι επόμενε εβδομάδε θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειε για να θέσουμε και να στέλνουμε τα σωστά μηνύματα. Έγιναν σωστέ προτάσει, τι οποίε καλούμαστε να συζητήσουμε. Να πω κατευθείαν για τη ζάχαρη. Στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο, υπερψηφίστηκε μια έκθεση με πλειοψηφία του 90% για να ολοκληρωθούν οι στόχοι αυτοί μέχρι το 2020 και αυτό το ψήφισαν όλες οι ομάδες. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτή την ε, πλειοψηφική θέση του Κοινοβουλίου και στο μέλλον. Ήταν λοιπόν ένα πρώτο βήμα, θα πρέπει να ακολουθήσει και το επόμενο τώρα, γιατί ξέρουμε ότι στο πρώτο βήμα αυτό κοιτάξαμε πιο πολύ το θέμα της σχέσης μεταξύ παραγωγού και μεταποιητή. Τώρα το θέμα είναι μεταξύ μεταποιητών και μεγάλων ομίλων και λιανεμπόρων. Στη Γερμανία ελέγχουμε ε, τι μερίδιο κατέχουν αυτοί οι μεγάλοι όμιλοι. Γι' αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί ακόμα η κατάσταση. Και ασκείται στους γεωργούς και στους, ε, στις αγροτικές ενώσεις μεγάλη πίεση ως προς τις τιμές. Κάτι άλλο τώρα που θα πρέπει να προσέξουμε το θέμα των πράξεων των εκτελεστικών. Διαβάζοντας τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέπουμε ότι παντού όλα ρυθμίζονται από εκτελεστικές πράξεις. Να προσέξουμε όμως, γιατί ως κοινοβούλιο θα πρέπει να διατηρήσουμε το πάνω χέρι και ιδιαίτερα ό,τι αφορά και το άρθρο 160, γιατί θα πρέπει να φροντίσουμε ως κοινοβούλιο όταν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, να μπορούμε να σταθούμε και στο ύψος των περιστάσεων σε ό,τι αφορά τις ευθύνε αυτές και όχι να βρεθούμε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τίποτα τελικά. Και πόσο σημαντικό είναι η κοινή οργάνωση αγοράς, το βλέπουμε και στον τομέα του βουτήρου, Διάβασα ότι δοκιμάζεται ο κλάδος αυτό στην Ευρώπη θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί και σωστά και γρήγορα ο τομέα αυτός, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ αργή η αντίδραση, η ανταπόκριση. Κάποιο άλλο πρόβλημα στην κοινή οργάνωση της αγοράς είναι η χρηματοδότηση των ε, ε, μέτρων για την αγορά. Δεν μπορούμε να φυλάξουμε μεγάλα ποσά για την αντιμετώπιση της κρίσης, ε, γιατί χρειάζεται πραγματικά δισεκατομμύρια και ασφαλώς ε, οι συνάδελφοι από τους άλλους κλάδους θέλουν και αυτή τα χρήματα αυτά. Χρειαζόμαστε ένα ποσό όμως το οποίο θα διατίθεται για τέτοιες κρίσεις στην αγορά και θα ήθελα να πω συνοψίζοντας ότι σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την ε, αγορά θα πρέπει να τους δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι πολύ βασικός παράγοντας για τη λειτουργία της του γεωργικού κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει λοιπόν όλες οι πληροφορίες ε, να συζητηθούν με τον εισηγητή του κ. Ταντάν και να ζητήσουμε σχετικές απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και νομίζω ότι έθιξες ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα το οποίο αφορά και όλους τους φακέλους σε ό,τι αφορά το πρώτο δεύτερο πυλώνα. Πρόκειται και το θέμα της εναρμόνισης με τη Λισαβόνα. Δεν καταφέραμε να βρούμε μια συμφωνία με την Πολωνική Προεδρία, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειες σε ό,τι αφορά τα θέματα χρηματοδότησης. Ε, αποτελεί μια βασική δυσκολία το ζήτημα αυτό, καθότι δεν υπάρχει συμφωνία. Ο Τζιωβάνι έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μισελ Νταντάν. Τον θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο με την έκθεση μου σχετικά με τα ανώτατα όρια πληρωμών. Είναι ένα θέμα που σχετίζεται με την ανάπτυξη της υπαίθρου και μας επαναφέρει στους κανονισμούς που ονομάζονται κανονισμοί ευθυγράμμισης. Ε, πρόκειται για την αυτόματη αποδέσμευση για τα ποσά στα πλαίσια της ανάπτυξης υπαίθρου. Θυμάστε ότι όταν συζητούσαμε εκείνους τους κανονισμούς εδώ στην Επιτροπή είχαμε εξετάσει το θέμα της αποδέσμευσης σε χώρες όπου είναι περιφερειοποιημένη η ανάπτυξη της υπαίθρου. Στην Επιτροπή λοιπόν είχαμε αναφέρει ότι για αυτές τις χώρες ε, είναι απαραίτητο να προβλέψουμε αποδέσμευση σε εθνικό επίπεδο αντισταθμίζοντας τις απώλειες μέσω των προγραμμάτων ανάπτυξης υπαίθρου. Αυτό το θέμα λοιπόν σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη υπαίθρου και εντάσσεται και στον οριζόντιο κανονισμό. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή έχω την πρόθεση να το κάνω, να ε, ρωτήσω τον κύριο Νταντά αν προτίθεται και εκείνος ε, να αναφερθεί στα όσα είχαμε αποφασίσει όταν κάναμε την ψηφοφορία για τον κανονισμό ευθυγράμμισης, διότι η αποδέσμευση θα πρέπει να προβλέπεται, ξαναλέω, σε εθνικό επίπεδο και για τα περιφερειακά Περιφερειοποιημένα συστήματα δεν ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια συστήματα αποδέσμευσης τοπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση όλων των κρατών μελών, ανεξάρτητα με το αν είναι περιφερειοποιημένη ή όχι η ανάπτυξη της υπαίθρου. Σας ευχαριστούμε. Τζοβάνι, Μπρίτα Ρέιμερς και ο κύριος Μποβέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Μισελ Νταντά για ε, την εξαιρετικά επικοδομητική προσέγγιση του καθ' όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Ε, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερος. Ο κύριος Νταντά υπογράμμισε ότι το παρελθόν είναι παρελθόν και δεν πρέπει συνέχεια ε, να αναμασούμε τα όλα όσα έχουν γίνει και μας μίλησε για... Και αυτό και για τις ποσοστώσεις. Θα πρέπει να είναι σαφές λοιπόν πότε πραγματικά λήγουν αυτές οι προθεσμίες και θα πρέπει να υπάρχει και ένα σαφές σχέδιο και για το πώς θα τερματιστούν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να τα αναβάλουμε όλα αυτά για την επόμενη αγροτική μεταρρύθμιση και να τα ξανασυζητήσουμε τότε. Αυτό ταλαιπωρεί και τους ε, γεωργούς αλλά και ουσιαστικά αναβάλλεται η συζήτηση. Χρειαζόμαστε ε, έναν απότερο στόχο και αυτό τι σημαίνει θα πρέπει να έχουμε και το θάρρος και την τόλμη να πούμε πού θα γίνουν αυτές οι περικοπές και πώς θα συνοδευτούν, από τι θα συνοδευτούν. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι φαίνεται ότι συμφωνούμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε επιστροφές για τις εξαγωγές ότι χρειαζόμαστε ιδιωτικά και δημόσια αποθέματα για να μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε σε περίπτωση κρίσης. Μια λύση της ανάγκης. Ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τις ε, ενώσεις παραγωγών θα πρέπει να προσέξουμε όμως γιατί αν τους απαλλάξουμε υπερβολικά από το δίκαιο του ανταγωνισμού μπορεί να αναπτυχθούν μονοπόλια. Και αυτό δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον των γεωργών να εξαναγκαστούν δηλαδή να συμμετάσχουν οι μη. Γιατί και πάλι θα είναι μονοπωλιακή η θέση που θα σχηματιστεί. Και αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι να προσέξουμε τι θα κάνουμε με τις πράξεις, τις επιλεκτικές και τις κατεξουσιοδότηση, γιατί ο σκεπτικισμός των πολιτών έχει να κάνει και λίγο με το πώς διαμορφώνεται μια κοινή κεντρική διοίκηση. γιατί δεν φοβάται ο κόσμος στο Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο και πολύ λυπάμαι αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς, ε, εσάς φοβάται το, ο κόσμος. Δεν έχετε διαφανείς δομές τις οποίες να μπορεί να καταλάβει ο πολίτης. Δεν καταλαβαίνει ο πολίτης πώς ε, καταλήγεται στις αποφάσεις που καταλήγεται και αυτό τον τρομάζει. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και είμαστε εμείς λοιπόν αυτοί που θα πρέπει να αποφασίζουμε σε περίπτωση που υπάρχει συναπόφαση και δεν νομίζω ότι θα καθυστερήσει αυτό τη διαδικασία γιατί ως τώρα τα πράγματα πάνε πιο γρήγορα στο Κοινοβούλιο από ό,τι στην Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να προσέξουμε αυτά που περιλαμβάνει η συνθήκη για τον πολίτη να τα τηρήσουμε. Ευχαριστώ. Ζωζέ Μποβέ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμμετάσχω κι εγώ στη συζήτηση για να συγχαρώ τον Μισελ Νταντάν για την εξαιρετική δουλειά του. Όντως πιστεύω ότι στα πλαίσια αυτού που του ζητήθηκε δύσκολα θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα πράγματα. Τα γενικά κεφάλαια νομίζω τα κάλυψαν οι συνάδελφοι με τα σχόλιά τους. Αυτά τα γενικά κεφάλαια μας προσφέρουν ένα γενικό πλαίσιο. Φυσικά ω προ τι λεπτομέρειες θα πρέπει να κάνουμε διευκρινήσεις μέσω των τροπολογιών φυσικά. Ω προ τι οργανώσεις ε, παραγωγών και τις διεπαγγελματικές ενώσει, ε, έχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία στην έκθεσή του κ. Ντάνταν σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει για τις Οργανώσει παραγωγών και το γάλα. Όντω, είναι ένα σύστημα που θα μπορούσε να επεκταθεί. Έχουμε δηλαδή παραδείγματα στο παρελθόν για το δίκαιο ανταγωνισμού. Όντω, ε, θα αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα, διότι δεν μπορούμε ταυτόχρονα να λέμε ότι δεν θέλουμε το κράτο να ελέγχει την ε, ε, παραγωγή και ούτε και θέλουμε να ελέγχονται οι διεπαγγελματικέ ενώσει, ούτε θέλουμε να ελέγχονται οι διενέξει ανάμεσα στου παραγωγού και τη μεταποιητική βιομηχανία. Τι θέλετε λοιπόν να επικρατήσει ο νόμο τη ζούγκλα, να το πούμε. Πάντως, σε επίπεδο κοινοβουλίου αρχίζουμε να ε, συντάσσουμε έναν οδικό χάρτη. Εγώ θα ήθελα να σας πω μόνο, απηχώντας την παρέμβαση της κυρίας Ρέιμερς, ε, το εξή: Όλοι μίλησαν για την ομαλή προσγείωση, το soft landing, σαν να είναι κάτι που θα έπρεπε να οργανώσουμε αφού μιλάμε για αεροπορία, γιατί δεν μιλάμε για απογείωση και μιλάμε για προσγείωση, γιατί όλο θέλουμε να προσγειωνόμαστε και να βγαίνουμε από ένα σύστημα. Είμαστε καινοτόμοι και απογειωθούμε για ε, τις νέες αγορές, τοπικές αγορές, ε, να ενισχύσουμε τη δράση μας για την περιφερειοποίηση, να, να μετεξελιχθεί δηλαδή το πλαίσιο της γεωργίας. Αυτό είναι καλή ιδέα κατά τη γνώμη μου τώρα. Ε, είμαστε δέσμοι του παλιού συστήματος να βρούμε την καλή φόρμουλα για το κρασί μέχρι να βγει από την ομάδα υψηλού επίπεδου γιατί ο στόχο είναι να καθυστερήσουμε. Λέτε εσείς 2030-2090. Οκ, okay, εγώ υπογράφω τώρα να κάνουμε τα ίδια και για το γάλα το 90. Καταπληκτική ημερομηνία, αλλά δεν μπορούμε να σοβαρευτούμε. Ας προσπαθήσουμε να επανασχεδιάσουμε με διαφορετικό τρόπο τη γεωργία και όχι να περιοριζόμαστε στα όσα έγιναν τη δεκαετία του 70 και του 80. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τον κύριο Μποβέ. Τελευταία παρέμβαση, κυρία Ντελάζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή ασφαλώς για την δουλειά που έχει κάνει. Να το ευχηθώ και κάθε επιτυχία για όλο τον όγκο της εργασίας που θα χρειαστεί να κάνει. Νομίζω ότι είναι η βασική έκθεση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον έναν πιο φιλελεύθερο κλάδο γεωργίας, το οποίο ασφαλώς δεν είναι αρνητικό αν ε, κάθε γεωργός ε, μπορέσει να έχει ένα εισόδημα, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα τόσο ιδανικός ο κόσμος και ξέρουμε όλοι ότι στο μέλλον θα έχουμε και διακυμάνσεις στον αγροτικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν μέσω από τις νομοθεσίες αυτές θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προβλέψεις για μια τέτοια κατάσταση. Αναρωτιέμαι λοιπόν ε, κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει πιο έντονη παρέμβαση και από την Επιτροπή Προϋπολογισμού κοιτάω και προς τον κύριο Λαβία μήπως θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν επαρκή κονδύλια για να μπορεί να γίνουν κάποια επιπλέον βήματα. Όταν για παράδειγμα υπερβούμε τους 30 ε, τόνους βούτυρος, να υπάρχει ένα σύστημα ε, πληστηριασμού σε ό,τι αφορά τώρα το πακέτο για τα γαλακτοκομικά. Νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο είτε μέσω των ευρωπαϊκών αρχών είτε μέσω των κρατικών αρχών μέσω του νομοθετικού πακέτου να παρέμβουμε στην ποιότητα, στην ποσότητα παραγωγής. Θα ορίσουμε την βιωσιμότητα μέσω αυτού του πακέτου, μέσω αυτού του μέσου. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό. Όλοι μιλάμε για τις χαμηλές τιμές του γάλακτος. Ε, Και αυτό θα ισχύει για όλες τις χώρες, αλλά φοβάμαι ότι αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη παραγωγή της Αμερικής και της ε, Νέας Ζηλανδίας. Άρα, το σύστημα αυτό το οποίο... Ένα σύστημα το οποίο θα περιορίσει τους παραγωγούς που μπορούν από ευρωπαϊκής άποψης να αγωνιστούν, θεωρώ ότι δεν είναι λογικό. Θα πρέπει λοιπόν να το ορίσουμε αυτό ε, μάλλον το προτινόμενο σύστημα ίσως να έχει κάποια λογική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο δεν ε, θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο να περιορίσουμε την παραγωγή, γιατί τελικά ουσιαστικά με ένα τέτοιο σύστημα πάντα είναι πίσω από την εποχή του. Έρχεται εκ των υστέρων. βλέπετε τη στιγμή που παίρνει απόφαση και λαμβάνει ένα μέτρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αλλάξει πάλι η κατάσταση στην αγορά για τις ποσοστώσεις στον ε, κλάδο της ζάχαρης. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η παρατηρήση της κυρίας Ράιμερς. Ας συμφωνήσουμε πότε θέλουμε να εκπνεύσουν τα συστήματα. Ίσως ε, να μην έχει έρθει η ώρα του συστήματος ποσόστοσης της ζάχαρης ε, για να καταργηθεί. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν συμφωνία για όλη την αλυσίδα της παραγωγής, για παράδειγμα, και με τους μεταποιητές της σάχαρης, για τη σοκολάτα για παράδειγμα, που περηφανεύονται ότι παράγουν με βιώσιμο τρόπο. Και τη στιγμή λοιπόν που θα συμφωνηθούν ε, το τι ακριβώς θα γίνει, τότε θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε και πότε θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που γίνεται και με τις ποσοστώσεις του γάλακτος, ένα οριζόντιο σύστημα κατάργησης. Ε αυτό που ισχύει δηλαδή στις ποσοστώσεις γάλακτος σήμερα. Ίσως να είναι χρήσιμο και για άλλους κλάδους παραγωγής. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε Έστερ, Ντελάνγκε, για την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να στείλει ένα μέλος. Ίσως λοιπόν αυτό θα μπορούσαμε να αποστέλουμε ένα μέλος για να εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε αυτές τις συναντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο αυτό, κύριε Νταντών, και αν δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι, ε, μετά από όλε αυτέ τι παρεμβάσει θέλω να κάνω δύο-τρει διευκρινήσει. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη διότι τα μπέρδεψα πριν με τι τρει εκθέσει που επανένταξα. Δεν είναι η έκθεση Ντόρφμαν, είναι Κάστρο για την ευθυγράμμιση. Και ακολούθησα απαρέγκλιδα όλες τις διατάξεις ε, περί ευθυγράμμισης για το δίκαιο ανταγωνισμού και για λόγους διαφάνειας ε, για τη σημερινή μας συζήτηση. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξή. Ε, είχα προβλέψει να πάρω διάφορου διάφορους από την ομολογία ή από τις κατευθυντήριες γραμμές. Όμως το άρθρο 103 της Συνθήκης Λισαβόνας δεν επιτρέπει παρέμβαση του Κοινοβουλίου για αυτά τα ζητήματα. Αποκλειστικά το Συμβούλιο μπορεί να κινηθεί βάσει πρόταση τη Επιτροπής και κατόπιν απλής νομοδότηση του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή λοιπόν θα καταθέσει προτάσει στο Συμβούλιο. Υπάρχουν και άλλα δύο σημεία για τα οποία πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε. Το θέμα της διαχείρισης ε, κινδύνου με το περίφημο κονδύλι για τη διαχείριση του κινδύνου που ε, δεν εντάσσεται στον προϋπολογισμό για τη Γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε αυτό το κονδύλι και δεν σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την έκθεσή μου, αλλά είναι ένα γενικότερο θέμα που απασχολεί ακόμα και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ελέγχου των προπολογισμών. γιατί υπάρχουν διάφορες σχολέ. πέρα από την ισορροπία που πρέπει να βρούμε ανάμεσα στου εισηγητέ, ούτω ή άλλω θα έχουμε τι τροπολογίε να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα. Ε, πιστεύω ότι ε, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε στο πεδίο εφαρμογή την ε, διάταξη περί επαγγελματικών ενώσεων. Είναι κάτι που λείπει σε σχέση με το ε, προηγούμενο σύστημα και που αντίθετα θα ήταν χρήσιμο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλου του συνεργάτε μου καθώ και τους σκιώδει. Πιστεύω ότι επικρατεί επικοδομητικό πνεύμα και θα κάνουμε πολύ καλή δουλειά και στο μέλλον. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Μισελ, εργάζεστε με εξαιρετικό τρόπο. Θα ήθελα να περάσω στο επόμενο σημείο. Τώρα ακολουθεί η παρουσίαση σε μιας μελέτης. Θα ήθελα όμω να υπενθυμίσω σε όλους του συντονιστέ, ε, ότι αμέσως μετά την μελέτη θα κάνουμε μια πάρα πολύ σύντομη σύσκεψη. Πιστεύω ότι σε μία ώρα θα έχουμε ε, τελειώσει. Μία ωρίτσα για να την παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε κατά τις 5.30 συνεδρία συντονιστών. Ε, ε, Έλεγα λοιπόν ότι θα ακούσουμε την ε, συγκριτική ανάλυση των επιδοτήσεων στον τομέα της γεωργίας ε, από τις βασικές εμπορευόμενες χώρες. Καλώς ορίσατε κύριε Ζαν Κρίστε Μπύρο από τη Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Πολιτικών καθώς και ο Ζαν Πιέρ Μπουτόν. ορίσατε. Θα σας δώσω αμέσως ε, το λόγο για να μας ε, παρουσιάσετε τις ε, επιπτώσεις των διαφόρων πολιτικών επιδοτήσεων. Παρουσιάστε την κατάσταση στον Καναδά, στην Ελβετία, κάνοντας την αντιπαραβολή με το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20 λεπτά κατανότα το όριο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε μία μελέτη η οποία αφορά τη σύγκριση της ε, γεωργικής στήριξης, της δημόσιας στήριξης της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλες χώρες. Υπάρχουν πολλοί ε, τρόποι στήριξης των γεωργών. Όταν γίνεται διεθνής σύγκριση πρέπει οι μέθοδοι να μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα είδη στήριξης. Παραδείγματος χάρη, αν δούμε τα στοιχεία τα οποία βλέπετε σε ένα, στο πρώτο γράφημα το οποίο έχετε λάβει, δηλαδή μέτρα στήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά ήδη. Μπορούμε να έχουμε τον κοινοτικό προπολογισμό, μπορούμε να έχουμε του εθνικού λογαριασμού, τα μικροοικονομικά δεδομένα και φτάνουμε σε εκτιμήσεις της τάξεως ε, των 50 δις ευρώ γεωργικής στήριξης. Αυτές οι πηγές συγκλίνουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αν προσθέσουμε τις ε, επιδοτήσεις ε, του ΩΣΑ, παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά τον άνθρακα, φτάνουμε σε υψηλότερα ποσά και αν προσθέσουμε και μια μορφή μεταφοράς που δεν είναι εμφανή στον περιορισμό, αλλά μεταφράζεται παραδείγματος χάρη ε, σε τιμές σταθερές, στηριγμένες, φτάνουμε σε ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Άρα η μεθοδολογία είναι αρκετά λεπτό θέμα, γιατί αν θέλουμε να συγκρίνουμε χώρες με διαφορετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που δίνουν συνήθω άμεσες ενισχύσεις και να τις συγκρίνουμε αυτές τις χώρες με χώρες που στηρίζουν τις τιμές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, μέτρα στήριξης τα οποία δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ εξετάσαμε εκ το σύναγγης αρκετούς δείκτες που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως είναι οι δείκτες του ΩΣΑ. Το PSE που είναι το ισοδύναμο της επιδότησης παραγωγού και τα ομαδοποιημένα ή γενικά μέτρα στήριξης που είναι τα μέτρα του ΠΟΕ. με μια αξία, θέλετε, νομική, γιατί πρέπει να σεβαστούν κάποια κατόφλια οι χώρες. Η στήριξη τώρα. Έχει μειωθεί το ποσοστό στις αναπτυγμένες χώρες, στις χώρες του ΟΣΑ και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε το μέσο όρο, ε, πολύ πιο υψηλά δηλαδή ε, σε σχέση με χώρες ε, όπως Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία. Πολύ πιο κάτω όμως σε σχέση με τη στήριξη που δίνεται στην Κορέα, την Ιαπωνία ή την Ελβετία. Προσεγγίζουμε το επίπεδο στήριξης όμως του Καναδά ή της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν με τον απλό αυτό σχετικά δείκτη βρίσκεται στο μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι εφ' εξής, η στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους γεωργούς είναι μια στήριξη κατά βάση ε, με άμεσες πληρωμές και όχι με τη στήριξη των τιμών. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον για τις παγκόσμιες αγορές, ότι δηλαδή η παρέμβαση έχει ως αποτέλεσμα πολύ λιγότερες διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές, ε, κάτι που ε, γίνεται ακόμη στη ΣΥΠΑ ή γινόταν στην Ευρώπη τη δεκαετία του 80. Σε σχέση με άλλες χώρες τώρα μπορούμε να πούμε πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παγκόσμιες αγορές έχει τρόπους στήριξης ε, που δεν θα ενοχλήσουν, αν θέλετε, τότε θα θίξουν πολύ άλλους παραγωγούς. Υπάρχουν χώρες για τις οποίες δεν ισχύει αυτό, όπως είναι αναδυόμενες κυρίως χώρες ή και η η Απονία, για να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Αυτό το γράφημα τώρα που βλέπετε δείχνει πώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τον καιρό προσεγγίσαμε τις τιμές ε, τους παραγωγούς με χωρίς τις, και βλέπετε τις παγκόσμιες τιμές ε, βλέπουμε να υπάρχει σύγκληση και αυτό είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ε, την αλλαγή της κοινή γεωργικής πολιτικής, όπου δίνεται λιγότερη βαρύτητα στους, μηχανικούς, στους μηχανισμούς παρέμβασης και στο τέλος της περίοδου βλέπουμε αύξηση ε, των παγκόσμιων τιμών. Βέβαια, το να μιλάει κανείς για τάση είναι ακόμα νωρίς, αλλά είναι κάτι εξαιοσημείωτο παρόλα αυτά. Βλέπουμε να υπάρχει λοιπόν μια αρκετά μεγάλη σύγκριση, δηλαδή ο λόγος προσεγγίζει το ένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, να δούμε τη στήριξη που δίνεται στις ΗΠΑ, Εκεί έχει παραμείνει αντικυκλική, πολύ πιο ασθενή στήριξη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό που βλέπουμε και πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι υπάρχουν στις ΗΠΑ μέσα εργαλεία που έχουν ως αποτέλεσμα ότι η στήριξη αυτή μπορεί να αυξηθεί πολύ, ιδίω ε, αν πέσουν οι παγκόσμιες τιμές. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα που παρέμεινε πολύ πιο κοντά ε, σε μια προστασία των ε, γεωργών από του αστάθμητου και απρόβλητου παράγοντε των αγορών σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια πιο ουδέτερη στήριξη σε σχέση με τι παγκόσμιε αγορέ, αλλά και σταθερότερη στήριξη. Σε κάποιες αναδυόμενες τώρα χώρες βλέπουμε ότι η γεωργική στήριξη έχει αυξηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για την Κίνα, για τη Βραζιλία ή για την Ρωσία. Για να κάνουμε λοιπόν αυτή τη διεθνή σύγκριση χρησιμοποίησαμε στοιχεία τα οποία συλλέγει κατά κύριο λόγο ο ΣΑ, αλλά είδαμε και επανεξετάσαμε με κριτικό μάτι και τη μεθοδολογία και έχουμε αλλάξει τους ε, δείκτες που χρησιμοποιεί ο ΣΑ. Ένα από τα προβλήματα με τους δείκτες αυτού, αυτούς είναι ότι είναι πάρα πολύ ε, ε από τις ε, διεθνείς διακυμάνσει. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς μετράμε το ισοδύναμο επιδότης παραγωγής παραγωγού. Αν το μετράμε σε δολάρια ή σε ευρώ, τα επίπεδα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Αλλά και οι τάσει μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν μια μεθοδολογία η οποία βασίζεται στην ε, ισοδυναμία της αγοραστικής δύναμης και λάβαμε υπόψη κατά τον τρόπο αυτό ότι με τη χειραγώγηση των σταλαγματικών ισοτιμιών ε, επηρεάζεται και η στήριξη στους παραγωγούς. Αυτό εξηγεί ιδίω ε, την μεγάλη στήριξη ε, στη Βραζιλία, την Κίνα και τη Ρωσία. Βλέπουμε εδώ για την περίοδο από το 95 έως το 97 στην Βραζιλία ότι φορολογούνταν οι γεωργοί στη Βραζιλία όπως στην Ουκρανία. Σήμερα όμως βλέπουμε σημαντικές ε, εξελίξεις, μεγαλύτερη στήριξη. Εάν λάβουμε υπόψη τώρα την πραγματική στήριξη λάβουμε υπόψη μας δηλαδή τις αλλαγματικές διακυμάνσεις ε, ιδιαίτερα, βλέπουμε ότι η Κίνα έχει αυξήσει πολύ σημαντικά τη στήριξή της. Η στήριξη της Γεωργίας σήμερα στην Κίνα σε πραγματική αξία υπερβαίνει συνδυασμένα τη στήριξη ε, τη γεωργική στις ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια πρέπει με επιφύλαξη να δούμε τα στοιχεία αυτά γιατί δεν είναι παγιωμένα, δεν είναι οπημένα τα στοιχεία του 10 ακόμα. Μπορεί να αλλάξει δηλαδή η κατάσταση, αλλά βλέπουμε αν επιβεβαιωθούν ότι υπάρχει πραγματική στήριξη στην Κίνα σε επίπεδα που αρχίζουν να είναι αρκετά πλέον υψηλά για την άμεση στήριξη των γεωργών, βλέπουμε τα ποσοστά στην Κίνα να προσεγγίσουν τα ευρωπαϊκά ποσοστά. Και αν λάβουμε υπόψη το σύνολο των επιπρόσθετων υπηρεσιών, επενδύσει για την έρευνα, για τι υποδομέ, βλέπουμε να προσεγγίσουν πολύ τα κινέζικα τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Αυτό το οποίο επίση είδαμε, και είναι, μια είναι ένα από τα συμπεράσματα τη μελέτη, είναι ότι η στήριξη, ε, τα μέτρα μάλλον στο πλαίσιο του ΠΟΕ, αυτό το aggregate measure of support, το γενικό μέτρο στήριξη. Σαστικά δεν έχει πια κάποιο νόημα αυτό το μέτρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε πάντοτε θετικά μέτρα στήριξης, ε, παραδείγματος χάρη για το σιτάρι. 100 ε, ευρώ τον τόνο, ακόμη και αν η παγκόσμια αγορά είναι στα 250 ευρώ. Ε, δεν υπάρχει δημόσια στήριξη της Γεωργίας βέβαια πια δεν είναι ενεργή αυτή, δεν ενεργός αυτή η τιμή, αλλά η μέθοδος του ΩΣΑ, με τη μέθοδο του ΩΣΑ, πάντοτε υπάρχει στήριξη με τον ΠΟΕ, συγγνώμη, μιλητής, γιατί βασίζεται σε ιστορικές αναφορές από τα τέλη της δεκαετίας του 80 με σύγκριση την τιμή στήριξη. Άρα δεν θεωρούμε ότι έχει πλέον και μεγάλο οικονομικό νόημα αυτό το μέτρο. Βέβαια εξακολουθούν τα μέτρα αυτά να είναι αρκετά χρήσιμα για να δούμε την ε, εξέλιξη της ιωρικής πολιτικής διαφόρων χωρών σε σχέση με τον ε, ΩΣΑ, αλλά δεν μπορούμε αυτό τον ε, δείκτη πλέον να τον χρησιμοποιήσουμε, αυτό το συνολικό μέτρο στήριξης. Επειδή είναι σημαντικό σε θέμα διεθνών δεσμεύσεων, βλέπουμε εδώ τις δεσμεύσεις απέναντι στον ΟΑΣΕ βλέπουμε ε, αυτό τη σύγχυση κόκκινες και μπλε ενισχύσεις, είμαστε πολύ πιο κάτω, στο 17% του κατοφλίου μας είμαστε. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως έχουμε περιθώρια λιγμών, σε περίπτωση που αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανασυνδέσει, όπως έγινε με το άρθρο 68, ένα μέρος των ενισχύσεών της. Επίσης αυξήθηκαν πολύ οι ενισχύσεις που δεν διαστρεβλώνουν την αγορά. Αυτό είναι το πράσινο τμήμα του γραφήματος. Ένα τελευταίο κομμάτι προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε την ευρωπαϊκή στήριξη με ορισμένες ε, χώρες στόχους για να δείξουμε αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα για την κοινή γεωργική και να δούμε εάν μπορούν να μας διαφωτίσουν οι συγκρίσεις αυτές. Είδαμε τη στήριξη κυρίως ε, στη ΣΥΠΑ. Όπως είπα είναι μια στήριξη που παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό αντικυκλική σε σχέση με την ευρωπαϊκή στήριξη που προστατεύει σε κάποιο βαθμό τους αγρότες από αντίξωες συνθήκες, αν είναι η ή αν οι τιμές δεν εξελίσσονται θετικά. Άρα ε, προσαρμογή. Και αν αυτή η στήριξη δεν είναι πολύ μεγάλη σήμερα, αυτό ισχύει, αυτό συμβαίνει γιατί είναι ε, υψηλέ οι τιμέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον στη συζήτηση που έχουμε σήμερα για το πώ μπορούμε να έχουμε πιο αντικυκλικές ευρωπαϊκές ενισχύσεις, γιατί αυτό φαίνεται ότι έχει κάτι θετικό, θα προστατεύσει από τις διακυμάνσεις ε, τους ε, αγρότες, να ψεκιμάσει τον τιμών και ταυτόχρονα οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις θέλουμε να είναι και πιο αποδεκτές από την κοινή γνώμη η οποία ε, εκπλήσεται όταν διαπιστώνει τα επίπεδα ε, ενιαίων πληρωμών. Σήμερα, ενώ είναι πολύ ψηλέ οι τιμέ αυτών των μεγάλων καλλιεργειών. Κατά την άποψή μα, παρά τα πλεονεκτήματα, αυτό το σύστημα των αντικυκλικών ενισχύσεων έχει και πολλά μειονεκτήματα και ιδίω ό,τι αφορά την ενδεχόμενη εφαρμογή του συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζουμε ότι είναι μια ε, καλή ιδέα. Δηλαδή το να είναι ο προϋπολογισμός συμβατός με το ευρωπαϊκό πλαίσιο στις ΗΠΑ μπορεί να αυξάνεται με κατά 10 δίσο ο προϋπολογισμός από τη μια χρονιά στην άλλη αν ε, πέσουν πάρα πολύ τιμές. Αυτό όμως φαίνεται πολύ δύσκολο να το χειριστεί κανείς στην Ευρώπη. Επίσης δείχνουμε, μάλλον στέλνουμε μηνύματα τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν ακριβώς ε, τα μικρά αποθεματικά. Και σίγουρα θα χρειαστεί ένα recoupling, μία σύνδεση με την παραγωγή. Επίσης δύσκολα καθίσταται αυτό συμβατό με την περιβαλλοντική αιρεσιμότητα και τους περιβαλλοντικούς όρους. Απ' την άλλη βέβαια μπορούμε να διαρωτηθούμε για το κατά πόσο είναι σκόπιμο να προσαρμόζει ένα Υπουργείο ε, τις ε, τιμές. Ενώ μπορεί να γίνει από τη μια χρονιά στην άλλη. Σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά βλέπουμε μια στήριξη η οποία όλο και περισσότερο επικεντρώνεται σε μέτρα διαχείρισης κινδύνων δεν θα επισέλθω ε, στην ανάλυση γιατί πριν από κάποια χρόνια κάναμε και μια σχετική ε, μελέτη. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι ότι τα ποσοστά αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, δηλαδή ε, ο λόγος του τι πληρώνει κατά φορολογούμενος και το τι παίρνει ο παραγωγός είναι μια χαμηλή αναλογία, χαμηλός λόγος. Άρα Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας γιατί με τις άμεσες ευρωπαϊκές πληρωμές αυτός ο λόγος είναι πολύ ψηλότερος. Αν δηλαδή θέλουμε να βοηθήσουμε τους γεωργού με αυτό το μηχανισμό, θα πρέπει να αυξήσουμε και τους προϋπολογισμούς, γιατί υπάρχουν περισσότερες απώλειες, διαρροές, ιδίως μέσω των συστημάτων των brokers, των μεσητών στις ΕΠΑ. Επίσης μελετήσαμε ιδιαίτερα την περίπτωση της Ελβετίας. Ε, πιστεύω ότι προχώρησε πιο πολύ τη μεταρρύθμιση που είχαμε και εμεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η περιβαλλοντική αρεσιμότητα έχει αναπτυχθεί περισσότερο και αυτό που είναι σημαντικό στην Ελβετία σε σχέση με την πρόταση τη Κομισιόν του Οκτωβρίου, ιδίω για το σκέλο του πρασινίσματο τη ΚΑΠ, και το Ecological Focus, την οικολογική εστίαση. Θα επεξεργαστούμε ακόμη το θέμα, αλλά από ό,τι βλέπουμε ε, στην Ελβετία... Τα μέτρα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στον τομέα της βιοποικιλότητας. Είναι η μόνη χώρα δηλαδή που φαίνεται να σημειώνει πρόοδο να περιορίζει την ε, υποβάθμιση της ε, βιοπικιλότητας. Έχουμε οικολογική εστίαση 7% και στις δύο περιπτώσεις, αλλά οι Ελβετοί παίρνουν και άλλα μέτρα συνδυασμένα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Έχουμε κάποιες προκατακτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τις επιφάνειες οικολογικού ενδιαφέροντος είναι διπλάσιες, 13-14%. παρότι σε ό,τι αφορά την παραγωγή θα έχει ε, ένα κόστος. Η Ελβετία δηλαδή είναι η μόνη χώρα όπου τα μέτρα για τη βιοπικιλότητα φαίνεται να αποδίδουν σε σχέση με τα γεωργοπεριβαλλοντικά ευρωπαϊκά μέτρα, τα οποία δεν έχουν πείσει μέχρι στιγμής ιδιαίτερα. Στο τελευταίο σκέλος ε, ασχοληθήκαμε με τις στρατηγικές των αναδυόμενων χωρών. Και εδώ ε, για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι η γεωργική στήριξη αυξάνεται, όπως είδαμε να συμβαίνει στην Κίνα και στη Ρωσία, λίγο στη, λιγότερο στη Βασιλεία, αλλά και στην Ουκρανία επίσης. Η στήριξη αυτή είναι προσανατολισμένη κυρίως στην παραγωγή για τα στρατηγικά ε, προϊόντα στην Κίνα, Στρατηγικά υπό την έννοια υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τους καταναλωτές και δεν θέλει η Κίνα να εισάγει για το ρύζι δεν έχουμε πολύ θετικέ εξελίξεις, αλλά για άλλα προϊόντα έχουμε. Επίσης ε, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις σε υπηρεσίες. Δηλαδή δεν ωφελούνται άμεσα η γεωργική παραγωγή, αλλά οι υποδομές σε πολύ μεγάλο βαθμό, κυρίως δε η έρευνα και η καινοτομία. Ο προϋπολογισμός στη Βραζιλία αυξάνεται με πολύ ταχύς ρυθμούς. Μιλάμε για αύξηση της ε, τάξεως πάνω από 20% ετησίως στη Βραζιλία για την έρευνα και την ε, καινοτομία. Αυτό το αναφέρει και η Κομισιόν στην πρότασή της. Νομίζω θα πρέπει να τα δούμε εκ παραλίλου. Ολοκληρώνοντας πάρα πολύ σύντομα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ε, το εισόδημα των γεωργικών παραγωγών. Οι ΕΠΑ προστατεύουν τους παραγωγούς από τις αντίξωες ε, συνθήκες και έχουν ε, μεγάλο προπλεξμό για την επισητιστική εθνική βοήθεια το 60% του γεωργικού προπλησμού τα λέγουμε food stamps. Στην Ελβετία, από την άλλη, βλέπουμε ότι στηρίζεται πολύ περισσότερο η παροχή των δημοσίων αγαθών. Η Κίνα στηρίζει την παραγωγή ειδικών συγκεκριμένων προϊόντων με στρατηγική προσέγγιση και στόχο την ε, επίτευξη οικονομιών, εξοικονόμηση πόρων και μεγιστοποίηση ε, των ε, εισαγωγών και οι αναδυόμενες χώρες εν γέννη, αλλά κυρίως η Βραζίλια και η Κίνα επενδύουν πάρα πολύ στο μέλλον μέσω της έρευνας και των υποδομών. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τους εμπειρογνώμονες. πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε και κυρίως αυτός ο τελευταίος πίνακας. Πολύ ωραία. Αρχίζουμε την ε, συζήτηση. Ο κύριος Ταραμπέλα, Μαγκίνε, Άγνιο, παρακαλώ. Μάρκ, ε, θέλω να ευχαριστήσω τον εμπειρογνώμονα για την παρουσίασή του, διότι Εντάξει, είναι προφανές ότι μπορούμε να το δούμε με την ησυχία μας, ε, όλη αυτή την έκθεση και την παρουσίαση, αλλά όταν ε, παρέπεμπε σε στοιχεία το ΩΣΑ, έχω την εντύπωση ότι δεν ε, λάμβανε υπόψη όλες τις επιδοτήσεις. Στην παρουσίασή σας όμως μας είπατε ότι παραδείγματο χάρη στη ΣΥΠΑ για το 2010 94 δις πήγαν στην επισητιστική συνδρομή. Ε, είναι σαφέστατο ότι κατά 94% πρόκειται για αγορά, εξαγορά εγχώρια παραγωγή από τι ίδιε τις είπα εννοώ. Για το 2010 ήταν τα στοιχεία, εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, ε, πρόκειται για επιδότηση. Πρέπει να συνυπολογιστεί και αυτή στις ε, επιδοτήσεις. Παρατηρείται επίση ε, ότι από πλευρά τη ε, Κίνα τη Βραζιλία και τη Ρωσία αυξάνεται η στήριξη προ τη Γεωργία και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια γεωργική στρατηγική που εστιάζεται γύρω από την ε, στήριξη τη παραγωγή. Εμεί είμαστε αφελεί εδώ, θέλουμε να επακούσουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, φτιάχνουμε τι επιδοτέ, αλλά τι αποσυνδέουμε μετά. Γιατί λοιπόν οι άλλοι όχι, ίσως αυτά που κηρύττουν στον ΠΟΕ δεν τα εφαρμόζουν στι χώρε του θα ήθελα λοιπόν πέρα από την παρουσίασή σας να μάθω το εξής. Έχουμε λάβει υπόψη όλες τις ε, επιδοτήσεις ε, για τη ΣΥΠΑ συγκεκριμένα, την επισητιστική συνδρομή. Ε, διότι ε, έχουμε ένα λόγο 1 προς 2,4 αν υπολογίζουμε τη στήριξη κατά κεφαλή ε, και, ή ανάλογα με τα τετραγωνικά χιλιόμετρα της έκτασης που μετρούμε. Δηλαδή, ε, δυόμιση φορές ε, μεγαλύτερη είναι η επιδότηση της ΕΠΑ σε σχέση με την Ευρώπη. Επίσης, μα μιλήσατε για τα αγροκαύσιμα και την ατέλειά τους, την εξαίρεση από την φορολογία. Ε, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε και δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στον γεωργικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να εξετάσουμε συνολικότερα τον προϋπολογισμό, ε, τον οποίο ένα τμήμα είναι η γεωργία, παρότι σε κάποιες χώρες αυξάνεται η στήριξη. Γι' αυτό σας είπα ότι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Νομίζω ότι άδικα νιώθουμε ένοχοι για τη γεωργία αν τα πάρουμε όλα αυτά υπόψη, μιλήσατε για τον αντικυκλικό χαρακτήρα της στήριξης ε, της παραγωγής, ε, ε, είναι σαφέστατο ότι για να βοηθήσουμε ε, τους ε, γεωργούς. Είναι πολύ πιο ευέλικτο το σύστημα όταν ε, αντισταθμίζουμε το εισόδημα όταν δεν επαρκούν αυτά που αποκομίζει από την αγορά. Θα ήθελα επίσης να εξετάσουμε όλους τους παράγοντες που δεν είναι γεωργικοί αμυγός και όλες οι επιδοτήσεις που δεν είναι γεωργικές αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζονται και θα ήθελα να ξέρω πού βασιστήκατε για τη μελέτη. Ευχαριστούμε Μάρκ, λέει ο Πρόεδρος. Ίσως αυτή η μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής ε, θα μπορούσε να είναι πιο προσαρμοσμένη στην ε, πραγματικότητα. Μαγκίνες, ευχαριστώ. Νομίζω ότι η τελευταία διαφάνεια είναι και πιο ενδιαφέρουσα. Όπου αναφέρεται ότι η Βραζιλία και η Κίνα επενδύουν στο μέλλον και αυτό συνεπάγεται ότι στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ που δεν επενδύουν θα υπάρξει αντίκτυπο. Θα μπορούσατε να κάνετε κάποια σχόλια, γιατί με εντυπωσίασε αυτή η διαφάνεια με τα πέντε σημεία αυτά. Θεωρώ ότι υπονοεί μία ανησυχία ότι η Ευρώπη δεν εξετάζει επαρκώς το μέλλον. Μιλήσαμε για την έρευνα και για τη μεταφορά γνώσης. Δώστε μας κάποια στοιχεία. Ένα σχόλιο το οποίο έγινε και ίσω δεν κατάλαβα λόγω τη μετάφραση. Υπάρχει ο κίνδυνο όταν λέμε ότι δεν υπάρχει δημόσιος, δημόσια υποστήριξη για τη χρηματοδότηση ε, για τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή είναι υψηλέ οι τιμέ. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τα εισοδήματα και υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των εισοδημάτων και των τιμών των, των ε, εμπορευμάτων. Σχολιάστε αν θέλετε και ύστερα σε ό,τι αφορά την Ελβετία είναι πραγματικά εντυπωσιακό το ότι γίνεται τόσα πολλά για την βιοποικιλότητα. Αν γίνεται το ίδιο, το οποίο δεν θα γίνει, δεν θα το επιτρέψει και η Επιτροπή μας, αλλά ποιος θα ήταν το κόστος και αντίκτυπος για την τιμή των τροφίμων. Και αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα στη τελευταία αυτή διαφάνεια είναι η γενικότερη κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες αγορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω και κάτι θετικό, έτσι, για αλλαγή. Ήταν πολύ καλή η παρουσίαση. Θα ήθελα και άλλα στοιχεία, όμως. Να σας στείλω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις, αν δεν σας πειράζει. Μιλώ στον κύριο που έκανε την παρουσίαση. Θα ήθελα και λίγο πιο πολλέ λεπτομέρειε. Θα σα αποστείλω λοιπόν γραπτά κάποιε ερωτήσει. ελπίζω να τι απαντήσετε. Με πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Κάπω έκπληξη μου, μου προκάλεσε το γεγονό ότι δεν αναφερθήκατε ιδιαίτερο στον Καναδά. Γιατί το είπατε ε, στην αρχή, το αναφέρατε. Είναι ενδιαφέρον το σύστημα που έχουν σε ό,τι αφορά την καλλιεργία, τις καλλιεργίες και την εκτροφή ε, βοηδών και των ε, φορολογικών κινήτρων. Δεν ξέρω αν αυτά συμπεριληφθήκαν απλά στην επισκόπησή σας, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά για το μεμονωμένο εκτροφέα καλλιεργητή. Αν ξέρει ότι επενδύοντας σε ένα μηχάνημα ε, μπορεί για παράδειγμα να έχει φορολογικό πλεονέκτημα και ανάλογα με τη χώρα του αυτό μπορεί να καθορίσει το κατά πόσο είναι ανταγωνιστικό ή όχι. Grazie ε, ευχαριστώ κύριος Ντες για να κλείσει. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και πραγματικά έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις να κάνω μιλώντας για τη ΣΥΠΑ και για την ε, λύση των αποζημιώσεων μέσω ασφάλειας για τέτοιες καταστροφές. Να σας ρωτήσω γιατί στην Αμερική Είναι εδώ και 40 χρόνια τόσο υψηλά, τόσο υψηλές αυτές οι αποζημιώσεις για α, φυσικές καταστροφές στις περιόδους περιόδες προεκλογικές. Τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτός ο τακτικός χαρακτήρας σε ό,τι αφορά τους ε, προϋποθέσεις του ΠΟΕ. Οι ΙΠΑ είναι αυτές που κρύβονται και συγχαίουν τις αγροτικές επιδοτήσεις με τις επιδοτήσεις για τρόφιμα. Ουσιαστικά αυτό ε, ενισχύει ιδιαίτερα την ε, Αμερικανική γεωργία. Τώρα σε ό,τι αφορά τους σχετικούς όρους. Κοιτώντας τι γίνεται για παράδειγμα στην Ευρώπη για τους όρους ε, σχετικά με το περιβάλλον. Υπάρχουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Καλιφόρνια. Αυτές οι, αυτές οι στρεβλώσεις λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. όταν πρόκειται για παραγωγή η οποία ε, προκαλεί, για παράδειγμα, ε, ζημιές στο περιβάλλον. Και σε ό,τι αφορά τις ε, ενισχύσεις αναγεωργό είναι πολύ πιο μεγάλες επιδοτήσεις αυτές στην Αμερική από ό,τι στην Ευρώπη. Δεκαπλάσιες, να σας πω. 17,5 στην ε, εκτάριο στην Ευρώπη 175 στην Αμερική ένα εκτάριο. Και συμφωνώ σε ό,τι αφορά αυτά που είπε η κυρία Μαγκίνες. Θα πρέπει να προσέξουμε χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ρωσία, όπου γίνονται προσπάθειες ε, να προετοιμαστεί για το μέλλον η γεωργία. Σε αυτές τις χώρες λοιπόν θα προσέξουμε, πρέπει να προσέξουμε πέρα από τις είπα. Grazie Albert. Adesso si Ευχαριστώ μου σε Ευχαριστώ. Με ικανοποίησε πάρα πολύ αυτή η παρουσίαση. Δεν μπόρεσα να την ακούσω εξ ολοκλήρου. Θα τη διαβάσω στη συνέχεια. Τέτοιες μελέτες έχουν ε, ιδιαίτερη αξία διότι μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργούν κάποια, συστήματα και να κοιτάξουμε, να στραφούμε προς το μέλλον της ε, κοινής γεωργικής πολιτικής. Ελπίζω οι συνάδελφοι από την... Ε, τα Υπουργεία Γεωργίας ε, στα κράτη-μέλη θα έχουν πρόσβαση επίσης σε τέτοιου είδους μελέτες. πιστεύω ότι το πρόβλημα ε, με την μεταρρύθμιση κοινή γεωργικής πολιτικής ε, είναι ότι δεν έχουμε μια ξεκάθαρη και ε, εικόνα ούτε και ανοιχτό πνεύμα σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας στον υπόλοιπο κόσμο. Εάν θέλετε μελλοντικά να έχετε δυνατότητα να εμπορεύεστε γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παγκόσμιες τάσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι χρηματοπιστωτικές αγορές τα εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της αγοράς σε όλες τις χώρες, αλλιώς δεν λειτουργεί συνολικότερα το σύστημα. Λοιπόν, αναλύοντας ε, όλα αυτά τα διαφορετικά παραδείγματα, τι πιστεύετε Πώς πρέπει να ε, χειριστεί τη μεταρρύθμιση κοινή γεωργικής πολιτικής η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ποιες χώρες ε, τόσο διαφορετικές εξάλλου μεταξύ τους θα μπορούσε να εμπνευστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. τα νέα εργαλεία της κοινή γεωργικής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρό μας. Θα ήθελα τώρα να ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονε μας ε, για να απαντήσουν στα πολυάριθμα ερωτήματα και να σα ευχαριστήσω εκ των προτέρων ε, για την παρουσία και για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ω προ το αν ε, συνυπολογίσαμε όλες τις επιδοτήσεις σα, απαντώ το εξή. Λαμβάνουμε υπόψη την επισητιστική βοήθεια, τον είπα, όμως ε, δεν λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό κονδύλι που διοχετεύεται στους ε, καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση στηρίζεται το εισόδημα των πολύ φτωχών ανθρώπων στη ΣΥΠΑ, αλλά ε, νομίζω ότι το αποτέλεσμα των νομισματικών μεταφορών στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αντίστοιχα αποτελέσματα. Όντως ε, είναι πολύ ψηλά τα μεγέθη και ξέρετε ότι έχει ληφθεί υπόψη αυτή η παράμετρο σε έναν από τους δείκτες ε, που χρησιμοποιήσαμε. Αυτό που δεν λάβαμε υπόψη είναι η βοήθεια μέσω των βιοκαυσίμων. Ούτω όσα αιτιολογίζει αυτές τις επιδοτήσεις με ε, ε, επιχειρηματολογία που ευσταθεί. Ισχυρίζεται ότι ε, δεν είναι ο πρωταρχικό στόχο η στήριξη του γεωργικού τομέα, είναι θέμα περιβάλλοντο και ενεργειακή ανεξαρτησία. Άρα δεν εντάσσεται πλήρω στο πλαίσιο τη κοινή γεωργική πολιτική ε, ο ΠΟΕ, ούτε και ο ΠΟΕ μάλλον, λαμβάνει υπόψη ε, αυτέ τι επιδοτήσει, διότι θεωρεί ότι έτσι αυξάνεται η παγκόσμια τιμή του η παγκόσμια τιμή των βιοκαυσίμων λόγω τη αύξηση τιμή του αραβό του παραδείγματο χάρη. Ε, γι' αυτό και, και δεν λάβαμε υπόψη αυτό το στοιχείο. Είναι σχετικά μεγάλο το πρόβλημα, διότι είτε μιλάμε για την Ευρώπη είτε για τη ΣΥΠΑ, είναι ε, ένας από τους βασικότερους τρόπους παρέμβασης για τους ελεούχους πόρους στην Ευρώπη και αντίστοιχα για τον αραβόσιτο ε, στις ΗΠΑ. Όταν ε, Κάνουμε τον υπολογισμό της ε, ε ισοδυναμίας, ε, λοιπόν, το έχουμε λάβει υπόψη, αλλά όχι σε σχέση με τους δείκτες ε, που χρησιμοποιήσαμε για τη μελέτη. Αν στην Ευρώπη, λοιπόν, έχουμε το 10% της φορολογικής ε, ελάφρυνσης για τα βιοκαύσιμα, σίγουρα η επιδότηση δεν είναι τόσο ισχυρή όπως τη είπα γιατί 40% της παραγωγής ε, του αραβόσιτου στη ΣΥΠΑ διοχετεύεται στην παραγωγή ε, βιοκαυσίμων. Η βασική επίπτωση δεν είναι η ατέλεια όπως σας έλεγα γιατί αυτό υπάρχει ακόμη αλλά κυρίως η υποχρεωτική ενσωμάτωση δηλαδή είναι ένα εργαλείο που δεν χρησιμοποιείται, δεν είναι μάλλον ένα δημοσιονομικό εργαλείο, είναι εργαλείο της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πέρα από τα βιοκαύσιμα όλες οι υπόλοιπε επιδοτήσεις είναι υπολογίζοντα Όταν σας μιλούσα για σημαντικό κόστος ε, μάλλον για ε, σημαντικές ε, μεταφορές, δεν, νομισματικές μεταφορές, δεν μιλούσα καθόλου για τα βιοκαύσιμα. Μιλάμε για το δεύτερο, δεύτερη ή τρίτη ε, θέση ε, στήριξη προ του γεωργού, στήριξη για τα ορυκτά καύσιμα, η οποία αντιβαίνει σε άλλε πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' αυτά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και στι νέε προτάσει. Για τον αντικυκλικό χαρακτήρα τη επιδότηση, δεν ξέρω αν ήμουν ξεκάθαρο στην παρουσίασή μου. Η άποψή μα. Ε, είναι μάλλον η εξή ότι αυτή η η επιδότηση δεν είναι προσαρμοσμένη στη, στα νέα δεδομένα. Αντίθετα με αυτά που κατάλαβε ο κύριος Ταραμπέλα, ούτως ή άλλως ε, στην τελική εκδοχή της έκθεσης θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Ω προ επενδύσει τώρα στον τομέα τη έρευνα ε, και τη σύγκριση ανάμεσα στην Ένωση και την ε, Βραζιλία, Έχουμε τις επενδύσεις ε, για την δημόσια παιδεία, τις επενδύσεις ε, για την έρευνα που λαμβάνονται υπόψη σε έναν από τους δείκτες που φέρει τα αρχικά TSE Πρόσφατα μας απασχόλησε αυτό το ζήτημα και τελικά το ποσό των δημοσίων επιδοτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν λάβουμε υπόψη και το 7ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο της έρευνας και τους διαφόρους οργανισμούς που ασχολούνται με την έρευνα, αν θυμάμαι καλά φτάνουμε στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Επιπροσθέτως έχουμε τα εθνικά κονδύλια και φυσικά οι ε, δαπάνες του ιδιωτικού τομέα για την έρευνα και την καινοτομία αλλά αυτό σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό της κοινή γεωργικής ε, πολιτικής ε, ε, δεν είναι σημαντικό μέγεθος. Τώρα, σε σχέση με την Ελβετία και την φαίνεται η πολιτική βιοπικιλότητα τη να είναι πιο αποτελεσματική από τα αγοροπεριβαλλοντικά έργα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστο παραγωγή δεν το έχουμε υπολογίσει ποσοτικά, διότι ε, ε, εκφεύγει, αν θέλετε, του πλαισίου τη ε, έκθεση. 6-7% τη καλλιεργήσιμη γη έχει η οικολογική εστίαση και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε όμω ότι θα αυξηθεί αναλογικά το κόστος ε, διότι έχουμε και το σύστημα της αγρανάπαυσης ε, όπου αφήνουμε ακαλλιέργητο η ε, στο ένα τμήμα και πιστεύω ότι η παραγωγή θα ε, μειωθεί κατά 3% το οποίο δεν είναι και αμεληταίο σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ρωτήσατε γιατί δεν αναφέρθηκα στον Καναδά. Ο Καναδάς λοιπόν στηρίζει εξίσου ε, τη Γεωργία όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ένας δείκτης που νομίζω είναι χαρακτηριστικός για το 2010 βλέπουμε ένα ποσοστό της τάξης του 20% η στήριξη βασίζεται σε ένα προϊόν, το γάλα για το υπόλοιπο υπάρχουν γεωργικές εγγυήσεις αλλά τίποτα παραπάνω. Πρόκειται λοιπόν ε, για ένα σύστημα εγγυημένης τιμής ε, μαζί με ποσοστώσεις ε, που αφορά μόνο τις δύο επαρχίες στην δύση του, στο δυτικό Καναδά. Το σύστημα αυτό μοιάζει με το αμερικανικό σύστημα, οπότε μπορείτε ε, όλες αυτές τις επικρίσεις που ενδεχομένως απευθύνεται στο αμερικανικό σύστημα να τις επεκτείνετε και στο καναδικό. Ως προς την ζημιά ε, του περιβάλλοντος, τις περιβαλλοντικές ζημιές ε, δεν έχουν υπολογιστεί, υπάρχουν Πολλοί άριθμα δημοσιεύματα σε επιστημονικές εφημερίδες ε, όπως ε, η Science εδώ ή και στη ΣΥΠΑ και βλέπουμε ότι η απώλεια της ε, βιοπικιλότητας, δηλαδή το κόστος της μείωσης του ποσοστού των νεκτερίδων που καταναλώνεται τα έντομα και άρα αυξάνεται η χρήση των εντομοκτώνων επειδή έχουμε λιγότερες νυχτερίδες και έχουμε και την μείωση Ε, της επικονίασης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στη Science πριν από τρεις μήνες είδαμε έκρηξη της ρήπανσης από αζωτούχα λοιπάσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οφείλεται καθαρά στη Γεωργία και έτσι δημιουργείται μια φιλοσοφικού τύπου ανησυχία. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι πρέπει να σταματήσουμε την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει κανένα νόημα, αλλά τέλος πάντων αυτά τα επιστημονικά στοιχεία είναι σχετικά πρόσφατα και εφόσον χρησιμοποιούσαμε στοιχεία του 2010 δεν αναφερθήκαμε σε αυτό στην έκθεση. Ε, τι άλλο να σας πω, οι λύσεις που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντας το παράδειγμα ε, κάποιων άλλων ε, χωρών. Κοιτάξτε, δεν είναι ο στόχος της έκθεσής μας. Η στήριξη προς ε, το εισόδημα ή η στήριξη της ε, παραγωγής. Αυτό είναι ένα βασικό δίλημα που πρέπει να μας απασχολήσει και το άλλο θέμα είναι αυτό του περιβάλλοντος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με άλλες νομοθετικές προτάσεις και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο ήδη από τον Οκτώβριο έχει επιληθεί του ζητήματος. Ευχαριστώ, θα περιοριστώ σε αυτά. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε μέσα στην έκθεση. Οφείλω να πω ότι Ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά τα στοιχεία. Στις 30 και 31 Μαΐου θα συνεδριάσουμε και πάλι. Λίγη συνεδρίασή μας τώρα και ζητώ από τους συντονιστές και τους εισηγητές να παραμείνουν, διότι θα κάνουμε